κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα υπερβούμε και τις δυσκολίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ζητήσω να μας δώσετε μία εγγύηση ότι θα αναζητήσετε μία λύση για την ενιακό και να μην υιοθετηθεί η πρόταση της Κομισιόν πριν να έχει βρεθεί μία λύση για όλα τα οριζόντια θέματα. Και πάλι ευχαριστώ Πρόεδρε και σας δίνω κατευθείαν το λόγο σας ευχαριστώ φυσικά για την παρουσία σας εδώ και για τη διαθεσιμότητά σας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο σε θέματα γεωργίας και ελίας. Η Πολωνική Προεδρία προσβλέπει σε καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των κοινωτικών θεσμικών οργάνων που θα γίνουν στο ίδιο ευχάριστο κλίμα. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία για πρώτη φορά αναλαμβάνει την ευθύνη άσκησης Προεδρίας στο Συμβούλιο και θέλουμε να αναμετρηθούμε με τον καλύτερο τρόπο με όλες τις προκλήσεις που συνεπιφέρει η άσκηση Προεδρίας στο Συμβούλιο. Η Πολωνία είναι μια μεγάλη χώρα με ανεπτυγμένο γεωργικό κλάδο. Γι' αυτό και το θέμα της γεωργίας, της ανάπτυξης υπαίθρου και της αλίας έχουν για την Πολωνία τεράστια σημασία. Τα γεωργικά ζητήματα αποτελούν προτεραιότητα της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Θέλουμε μια ασφαλή Ευρώπη για, στα τρόφιμα, την ενέργεια και την άμυνα. Στα πλαίσια αυτά, η Πολωνία θέλει να επισημάνει την θεμελιώδη σημασία που έχει η επιστημιστική ασφάλεια για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, ιδιαίτερες ε, λειτουργίες που θα επιτελέσει η μεταρρυθμισμένη, και το τονίζω, η μεταρρυθμισμένη γεωργική πολιτική. Στα πλαίσια γεωργία και ανάπτυξη υπαίθρου, η Πολωνική Προεδρία θα επικεντρωθεί κυρίω στη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Επιπλέον, σημαντικό ε, ε, τομέα συζήτηση θα είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στην Ήπεθρο. Ε, θέλουμε να προκαλέσουμε πραγματικά διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της γεωργίας και ταυτόχρονα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικό στοιχείο της κοινή γεωργικής πολιτικής που συνδέεται με την πολιτική συνοχή αλλά και την ενεργειακή μας πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, είναι θέμα τεράστιας σημασίας για την Πολωνική Προεδρία. Ε, το θέμα αυτό αποτελεί εδώ και πολύ καιρό αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων στα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Και μάλιστα συζητήθηκε πρόσφατα η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική μέχρι το 2020. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ανακοίνωσης που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα. Κεντρικά ζητήματα που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα που συζητήθηκαν και στο Συμβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο θέλουν να συνεχίσουν την επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το νομοθετικό πακέτο, η Πολωνική Προεδρία σκοπεύει ήδη από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει εντατικές συζητήσεις και στο Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, θα είναι η πρώτη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα καλύπτει 27 χώρες μέλη. Θα είναι ταυτόχρονα και η πρώτη μεταρρύθμιση που θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που είναι τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής. Αναφυσβήτητα και τα δύο θεσμικά όργανα θα πρέπει να λάβουν υπόψη το υπέρτερο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας προκειμένου να καταλήξουν σε συμβιβασμούς και συμφωνίες. Οι μέχρι τώρα εργασίες δείχνουν ότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής θα καθοριστεί από κοινού με τις εργασίες για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως μας υπενθυμίσατε πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό και η Πολωνική Προεδρία έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες για τον προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο κρίνει ότι η δική σας Επιτροπή, αλλά και η Ειδική Επιτροπή ΣΟΥΡΕ για τις πολιτικές προκλήσεις και τους, δημο, τους δημοσιονομικούς πόρους, θεωρούν ότι και μετά το 2013 θα πρέπει να διατηρηθεί το ισχύον επίπεδο χρηματοδότησης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις συζητήσεις ε, για πραγματικά εμβριθείς αλλαγές στην κοινή γεωρική πολιτική που θα οδηγήσουν σε μια απλούστευση ξεχνώντας τους ε, ιστορικούς ε, τίτλους και τα σημεία αναφοράς και θεσπίζοντας νέα και αντικειμενικά κριτήρια αποδεσμευόμενοι από τα ιστορικά σημεία αναφορά και με νέα αντικειμενικά κριτήρια. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια κοινή γεωρική πολιτική που θα είναι δίκαιη, θα προσανατολίζεται στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κοινό στόχο και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, το γύρο της Δόχα, τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Μερκοσούρ, και τις συζητήσεις σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις, ιδιαίτερα στη ΦΑΟ, στην ομάδα G20 και στον Κόντεξ Αλιμεντάριους. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τις απόψεις της Πολωνικής Προεδρίας για ορισμένες, αυτέ από αυτές τις διεθνείς διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το γύρο της Δόχα, μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο προσβλέπει σε διαθέτηση των μεμονωμένων ε, ε, εγχειρημάτων. Και μετά από τις, την πρώτη σοδιά για τα λιγότερα επίμαχα ζητήματα, Κατά τη γνώμη της Προεδρίας, η πρώτη αυτή σοδιά δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και στις διαπραγματεύσεις για το Μερκοσούρ Όλες οι προσφορές της Ευρωπαϊκής Προεδρίας θα πρέπει να τηρήσουν την διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τελευταίες ε, ειδήσει που έχουμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου δείχνουν πού βρίσκονται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών. Θα πρέπει εκ του να παρακολουθούμε την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη ΦΑΟ, η Πολωνική Προεδρία στηρίζει την δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξασφάλιση διεθνού και συντονισμένη απάντηση στο πρόβλημα τη έλλειψη τη επισητιστικής ασφάλεια. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από πείνα ή υποσυτισμό. Είναι μια σημαντική πρόκληση λοιπόν αυτό και για την Ευρώπη. Οι εργασίες και στο G20 υπό την Προεδρία της Γαλλίας έχουν τεράστια σημασία. Η Προεδρία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την απαραίτητη συνέχιση των υπουργικών συσκέψεων του G20 του προηγούμενου μήμα και τα θέματα της, του προγράμματος εργασιών σε ό,τι αφορά τη Διακύμαση των τιμών τροφίμων και του γεωργικού εμπορίου. Θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχει η Επιτροπή του Κόντεξ Αλιμεντάριους, ΦΑΟΠΟΕ, ε, γιατί καθορίζει τις ε, διεθνείς προδιαγραφές στα πλαίσια του κοινού προγράμματος προδιαγραφών τροφίμων της ΦΑΟ και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Οι κανόνες αυτές ε, αποτελούν σημείο αναφοράς και στην ΠΟΕ σε περίπτωση διαφορών που αφορούν τη συμφωνία για τη χρήση υγειονομικών ή φυτοϊγειονομικών μέσων στα πλαίσια της ασφάλειας των τροφίμων. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στα πλαίσια της Πολωνικής Προεδρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του Κόντεξ Ανιλιμεντάριους και μάλιστα θα έχουμε σύντομα τρεις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής της, ε, του Κόντεξ Αλιμεντάριους που θα αφορούν τον έλεγχο εισαγωγή και εξαγωγή των διαφόρων, συστημάτων, ε, των διαφόρων τροφίμων και το σύστημα πιστοποίηση. και μάλιστα τα τρόφιμα ε, τρόφιμα ιδιαίτερη διατροφική σημασία καθώ και την υγιεινή των τροφίμων. Θα ήθελα εν συντομία τώρα να σα παρουσιάσω τη θέση τη Πολωνική Προεδρία για διάφορα άλλα θέματα που ήδη συζητούνται στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και θα απασχολήσουν και την ε, Επιτροπή. Ξεκινώ από το πακέτο για την ποιότητα των τροφίμων. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο ποιότητας που απαρτίζεται από δύο προτάσεις. Η πρώτη αφορά το σύστημα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και η δεύτερη τροποποιεί τους ισχύοντες κανόνες ε, εμπορίου για τα γεωργικά προϊόντα. Τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, σημείωσαν σημαντική πρόοδο ό,τι φορά την μελέτη αυτών των δύο προτάσεων. Βέβαια, ε, εκκρεμούν και κάποια θέματα που χρήζουν πολιτικής απόφασης. Το Συμβούλιο προσβλέπει σε τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά η Πολωνική Προεδρία θα φροντίσει να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές για όλους λύσεις. Σε ό,τι αφορά το πακέτο για το γαλακτοκομικό τομέα, η Προεδρία θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή, τον κύριο Νίκολσον, σε ό,τι αφορά την ε, εξασφάλιση των κατάλληλων ε, μέτρων για τον τομέα αυτό, γιατί η πρόσφατη κρίση, μάλλον η κρίση του γαλακτοκομικού τομέα του 2008, καθιστά επιτακτική ανάγκη τη λήψη τέτοιων μέτρων και δραστηριοτήτων για να εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον για τους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά το θέμα τη ε, ταυτοποίηση των βοηδών, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ε, προτάσεις για μέτρα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των βοηδών, απλουστεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Είμαι πεπισμένο ότι και η δική σας Επιτροπή θα είναι ανοιχτή για να εξετάσει οποιοδήποτε μέτρο που στόχο έχει τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους για τους γεωργούς αλλά και για τις τοπικές και εθνικές αρχές. Το ίδιο ανοιχτό θα είναι και το Συμβούλιο και μάλιστα εμείς ε, θέλουμε το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσουμε την ε, εξέταση αυτών των προτάσεων έχοντας υπόψη την ανάγκη ε, επικοδομητικής συνεργασίας με την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και μάλιστα πριν τα τέλη του έτους. Επόμενο ζήτημα που είναι σημαντικό και για το, και για Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι το θέμα της ευημερία των ζώων. Ελπίζουμε το φθινόπωρο του έτους αυτού να υποβάλει την πρότασή της ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό 1 του 2005 σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Έρχομαι τώρα σε κάποια φυτογειονομικά θέματα. Οι πρώτες διατάξεις, οι φυτογειονομικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίστηκαν πριν από 30 χρόνια περίπου. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει αλλάξει. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση αυτών των κανόνων είναι απαραίτητη. Η παγκοσμιοποίηση και οι κλιματικές αλλαγές αυξάνω τον κίνδυνο της μετάδοσης των νόσων και των παρασιτών και παθογόνων παραγόντων. Αυτό επηρεάζει και το γεωργικό κλάδο αλλά και το περιβάλλον. Επίσης ε, είναι επιτακτική ανάγκη ο εξυγχρονισμός και η απλούστευση της ε, σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας ό,τι αφορά την εμπορία των σπόρων και του υλικού διάδοσης φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια εναρμονισμένη και ανταγωνιστική ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά την υψηλή ποιότητα των σπόρων και του υλικού πολλαπλασιασμού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να λάβουμε υπόψη την όλο και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση και τις διεθνείς προδιαγραφές. Και στους δύο αυτούς τομείς η Πολωνική Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ολοκληρώσει κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες με βάση τις νομοθετικές προτάσεις. Και μάλιστα θα ξεκινήσουν και οι δημόσιες συζητήσεις στο Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική προώθηση. Η πράσινη βίβλο δημιουργεί την ε, ευκαιρία ε, διαμόρφωσης μιας κοινή αντίληψης για έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την προώθηση και την πραγματοποίηση των κοινών στόχων της πολιτικής προώθησης. Το θέμα της πρόθεσης θα αποτελέσει σημαντικό θέμα στο άτυπο συνέδριο, το Υπουργικό Συνέδριο που θα γίνει στο Βρότσοφ τον Σεπτέμβριο. Θα ήθελα τέλος να πω λίγα λόγια για την προσαρμογή της γερικής νομοθεσίας στη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι τεχνικές εργασίες και κυρίως τέσσερα σημαντικά νομοθετικά εργαλεία σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή ο κανονισμός για τις άμεσε πληρωμέ, ο κανονισμός για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς, ο κανονισμός ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ο κανονισμός για τη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, οι εργασίες για αυτούς τους ε, κανονισμούς βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Σε ό,τι αφορά ορισμένα έγγραφα, ήδη έχουν ξεκινήσει τριμερείς επαφές και με τόσο λίγο θα ξεκινήσουν και για τα υπόλοιπα έγγραφα. Με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε την πληροφορία ότι για τα θέματα αυτά και εσείς προσωπικά κύριε Πρόεδρε δεσμευθήκατε να συντονίσετε τις συζητήσεις ό,τι αφορά αυτά τα τρία μείζωνα νομοθετικά κείμενα. Και μάλιστα χαιρόμαστε και εμείς με τον στόχο αυτό να διεκπαιρώσουμε όσο το συντομότερο γίνεται αυτές τις αποφάσεις, χωρίς όμως να επιβαρύνουμε υπερβολικά τη συζήτηση για την κοινή γεωρική πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου με τη διαβεβαίωση ότι η Πολωνική Προεδρία το επόμενο εξάμεινο δεν θα αφιστεί προσπαθειών προκειμένου να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων κάτι που θα δημιουργήσει στέρεες βάσεις για φιλόδοξες και ισορροπημένες συμφωνίες στο δεύτερο εξάμεινο του 2011, αλλά φυσικά και αργότερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρεκ, ευχαριστώ για την παρέμβασή σου, ευχαριστώ για τη δέσμευση της Πολωνικής Προεδρίας και ευχαριστώ και για την τακτική σου παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και στην Ολομέλεια, την περίσμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ε, σας ε, είχαμε και Πραγματικά έχουμε 6 μήνες εντατική εργασίας μπροστά μου και φυσικά αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο στα νομοθετικά μα καθήκοντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Λοιπόν, όποιο ζητήσει το λόγο μπορεί να πάρει το λόγο αμέσω. Σας ε, καταρχήν. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Νομίζω πως από τη σκοπιά του ΕΛ και η έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια των τροφίμων και νομίζω πως όλοι στην Επιτροπή μας συμφωνούν με αυτή την ε, ανησυχία που αναφέρατε. Είναι νομίζω η βασική ανησυχία όλων μας. Ανησυχία όλος ο κόσμος και θα πρέπει να είναι και πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα σας στηρίξουμε στις ε, προσπάθειές σας να έχετε αυτό ως προτεραιότητα. Και βεβαίω ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο τη μεταρρύθμισης τη γεωργική πολιτική. Αναφέρατε τον προπολογισμό, τεράστια ανησυχία και εμεί θέλουμε να διατηρηθεί τουλάχιστον ο προπολογισμό στο τωρινό του επίπεδο. Ένα ερώτημα έχω για τη μεταρρύθμιση. Έγινε αναφορά στην έβρεση νέων κριτηρίων και βεβαίως ε, όλοι προσπαθούμε να γίνει κάτι τέτοιο με μια ρεαλιστική προσέγγιση. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορείτε να μας πείτε σήμερα ε, ως προς αυτό δεδομένων των ανησυχιών που έχουμε για δικαιοσύνη, όσον αφορά την ε, πολιτική αυτή, το να διατηρηθεί επίσης η παραγωγή τροφίμων σε όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίω τα περιφερειακά ζητήματα που αφορούν την γεωργική πολιτική. Κάτι που σχετίζεται με αυτό αλλά δεν αναφέρατε και ίσως θα θέλατε να το κάνετε. Η Κομισιόν έχει εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά το ποσοστό της τιμής καταναλωτή που καρπώνεται ο παραγωγός, δηλαδή το πώς δουλεύει όλη αυτή η αλυσίδα. Εμείς πιστεύουμε πως καμιά φορά αυτό λειτουργεί εις βάρος των παραγωγών και αγροτών και τι θα μπορούσε να κάνει η Προεδρία σας γι' αυτό για να υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη στην ε, αλυσίδα παροχής ε, τροφίμων γιατί θεωρώ πως υπάρχει μια ανισορροπία δυνάμεων αν θέλετε και κάποιοι άλλοι εκτός από τους αγρότες εμποφελούνται και βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα με αυτό. Επίσης, σχετικό, ο τομέας των γαλακτοκομικών που απασχόλησε και την έκθεση Νίκολσον. Υπάρχουν ανησυχίες στα κράτη-μέλη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την εποχή μετά τις ποσοστώσεις γάλακτος και πρέπει κάτι να υπάρξει ως κατεύθυνση για τους παραγωγούς και είναι νομίζω ένα σημαντικό θέμα. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για τα κράτη-μέλη εκείνα όπου ήδη υπάρχουν δυσκολίες από τις ε, ποσοστώσεις και το τι θα γίνει εντός του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν. Βεβαίω σημαντικό και αυτό το οποίο είπατε για, την ανανεώσιμη, για τις ανανεώσιμες υγιές ενέργειες, χωρίς να επηρεάσουμε την ασφάλεια των τροφίμων, ε, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο νομίζω για εμάς αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να περάσω τώρα στην εμπορική πολιτική, γιατί είναι κάτι που απασχολεί γενικά την Προεδρία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι σκόπευτε να κάνετε για τις συμφωνίες με το Μερκοσούρ. Εμείς στην Επιτροπή μας, το ΕΛΚ, ανησυχούμε για ασυνέπειες στην εμπορική πολιτική. Προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τη γεωργική πολιτική, να πείσουμε και τους αγρότες αλλά βλέπουμε από την ε, πλευρά του εμπορίου κάποια βήματα που θα φέρουν σε μειονεκτική θέση την γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ρωτήσω πώς ε, θεωρείτε πως θεωρειτε πως μπορουν να συμβιβαστούν αυτές οι δύο πολιτικές και όχι να αποκλίνουν. Όσον αφορά τις προδιαγραφές, πράγματι έχουμε γεωργούς που καλλιεργούν με υψηλές προδιαγραφές, αλλά τι σημαίνει αυτό πάντα με τις αγωγές από τρίτες χώρες. Αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο ερώτημα. Έχουμε διμερείς συμφωνίες που προωθούνται και συμφωνίες ε, του ΠΟΕ. Και η ανησυχία μου είναι πως ε, θα υποχωρήσουμε πάρα πολλές φορές ε, στο εμπόριο και θα έχουμε πολλά μειονεκτήματα στην γεωργία και θα έχουμε προβλήματα ασφάλειας τροφίμων. Θα ήθελα να το μεταφέρετε αυτό στο Συμβούλιο και να μας απαντήσετε όταν θα επανέλθετε για το ζήτημα της εμπορικής πολιτικής. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, για την ευζοία των ζώων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το δείτε αυτό ως εξή. Ας δούμε την ύπαρξη νομοθεσία και να την εφαρμόσουμε πλήρως. Υπάρχει πάντα μια ανησυχία πως συσσωρεύεται η νομοθεσία και δεν εφαρμόζουμε την υφιστάμενη. Οπότε σας παρακαλώ να εφαρμόσετε πλήρως αυτά τα οποία ισχύουν και να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες που υπάρχουν εδώ μέσα για τον τομέα της παραγωγής αυγών για τα πουλερικά σε συστοιχίες γιατί αντιμετωπίζουμε βεβαίω κάποιε συνέπειε, Πολλοί παραγωγοί δεν είναι έτοιμοι, κάποιοι άλλοι είναι. Πρέπει να δούμε πώ θα εφαρμοστεί δίκαια αυτή η νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα έχει μεγάλη σημασία. Αναφέρατε το πακέτο ποιότητα των τροφίμων. Ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σα, νομίζω μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά το γενικότερο μήνυμα είναι πως η Ευρώπη θα πρέπει να είναι συνεπής σε σχέση με αυτά τα οποία λέει ε, για τη γεωργία και με αυτά τα οποία κάνει στο εμπόριο. Εγώ δεν βλέπω κάποια συνέπεια εδώ πέρα. Δεν βλέπω τον ε, Επίτροπο Εμπορίου να μιλάει τόσο ξεκάθαρα όσο η αρμόδια για τη Γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να είστε ειλικρινεί και να θίξετε το θέμα σε υψηλό επίπεδο. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία καθώς αναλαμβάνεται αυτή τη μεγάλη πρόκληση της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Γκαρσία Περάς παρακαλώ. Και κατόπιν του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για τις εργασίες σας στο επόμενο εξάμεινο, γιατί ε, χωρίς ε, καμία αμφιβολία το δικό σας έργο θα είναι και δικό μας ε, και αν πετύχετε θα είναι και δική μας επιτυχία και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ε, σε ό,τι αφορά το μέλλον της ΚΑΠ και το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ε, σημαδέψουν το μέλλον της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση για τη δεσμή για την ποιότητα καθώς είμαι εισηγήτρια. Να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε Ξέρετε ότι είχαμε κάποιες συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η Επιτροπή ήδη στη θέση που έλαβε τόσο για τον κανονισμό για τα καθεστώτα ποιότητα ε, όσο και για τα πρότυπα εμπορίας ε, και μπορούμε να καλέσουμε την ε, Πολωνική Προεδρία να λάβει υπόψη αυτή την θέση απέναντι στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένα δύσκολα θέματα που πρέπει να προσεγγιστούν αλλά νομίζω ότι αυτό το κοινοβούλιο ε, παρόλο που έχει αποκλίνουσες απόψεις μπορούσε να καταλήξει σε ένα γενικό πλαίσιο με ευρία πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρχει και καμία αμφιβολία ότι και το Συμβούλιο μπορεί να ακολουθήσει την ίδια αυτή γραμμή και να συνεργαστεί έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου ε, να έρθει στο φως αυτό το νομοθετικό πακέτο. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την ποιότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και να ε, δημιουργήσουμε αυτή την προσθεμένη αξία των προϊόντων μας ε, και να σημειώσουμε πρόοδο σε όλες τις πολιτικές που αφορούν την πρόθεση των ε, αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω αυτή τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία και ελπίζουμε τα αποτελέσματα να είναι θετικά για το καλό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ροντούστο και κατόπιν καλνιέται. Entschuldigung, Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το όνομά μου. Ε, είναι η προφορά. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι για το ότι είστε εδώ. Σας άκουσα προσεκτικά. Αλλά άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τους Γερμανούς αγρότες στο Κόμπλεντ, στην ε, συνάντηση των Γερμανών αγροτών και εκεί πέρα μου είπαν πως ε, θεωρείτε πως ε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ άδικη η κατανομή των άμεσων πληρωμών. Μιλήσατε τώρα μόλις ε, για νέα αντικειμενικά κριτήρια και κατάργηση των παλαιών. Μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ τι εννοείτε εδώ πέρα συγκεκριμένα και τι θα προτείνετε για το τι θα πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες από εσά μετά. Είπατε πάλι στην ημέρα των αγορτών πως οι ποσοστώσεις για το γάλα θα εξαντληθούν το 2015 και θεωρείται αυτό πάρα πολύ προβληματικό. Εκεί πέρα είπατε πως ήταν μεταφραστικό λάθος αλλά δεν ήμουν τόσο σίγουρη και μια που είστε εδώ πέρα σήμερα θέλω να μας ε, πείτε. Θέλετε να καταργήσετε τις ποσοστώσεις ή θεωρείτε πως πρέπει να διατηρηθούν. Έχετε δίκιο πράγματι πως πρέπει να αναπτύξουμε άλλα μέσα για τις ε, μικρές επιχειρήσεις για να μην καταστραφούν, αλλά το θέμα δεν είναι η δική μου άποψη, αλλά η δική σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ε, Πολωνική Προεδρία γιατί δεν είναι, δεν είναι εύκολα αυτά τα οποία έχετε να κάνετε αλλά εμείς θα σας στηρίξουμε και θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί υπάρχουν ε, ζητήματα στα οποία οι θέσεις μας ε, ταυτίζονται, δηλαδή τα αντικειμενικά κριτήρια στα οποία πρέπει να βασιστεί η κοινή γεωργική πολιτική. Επίσης εκτιμώ την ε, θέση σας ε, για το πολιετές πλαίσιο για ζητήματα που πρέπει να επιληθούν όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω για τη θέση των αγροτών στη Λετωνία, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι από τις προτάσεις της Κομισιόν. Στη Λετωνία έχουμε τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές, 94 ευρώ ανά εκτάριο. Και το 2020, 20 χρόνια μετά την εξαρτησία, θα λαμβάνουμε 144 ευρώ ανά εκτάριο. Μόλις πάνω από το μισό της μέσης ε, πληρωμής ανά εκτάριο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν πως αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν δεν είναι ευθυγραμμισμένο με αυτό το οποίο έχει πει η ίδια η Επιτροπή. Πως ε, δηλαδή θα είναι δίκαιη και ισορροπημένη η στήριξη των γεωργών. Και μας έχετε πει πως ε, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνει ένα ποσό αναλογικό και θα πρέπει να υπάρχει και ένα πλαφόν. Οπότε εγώ θεωρώ πως κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να βάλει λιγότερο από 80% και περισσότερο από 120% των μέσων πληρωμών στην Ένωση. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη πως ε, τα κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν ε, πολύ λιγότερο από το 50% της μέσης πληρωμής ε, έχουν πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει το στομότερο δυνατόν το 2014 δηλαδή η εξορρόψη αυτή και να μην ε, διαρκέσει αυτή η περίοδος περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και μπορείτε να βασίζετε σε μας για την στήριξη μας. Ευχαριστώ, Ντόρφμαν και Κατοπιλιάρ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και κάνετε αυτή τη συζήτηση μαζί μας. Θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Κανιέτε για την κατανομή των άμεσων πληρωμών γιατί ξέρετε πως εμείς ε, ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Κάποιοι την θεωρούν δίκαια, κάποιοι άδικοι, αλλά δεν μιλάμε για το τι συμβαίνει εντός των κρατών μελών. Αναφέρω τη δική μου περιφέρεια, παραδείγματος χάρη, η η γειτονική περιοχή ξέρετε πως ε, η κατανομή μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα είναι 1 προς 10 και η ιστορική σύνδεση με την ε, παραγωγή έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ, σε στο να ευνοείται αυτή η περιοχή σε σχέση με άλλες ε, πιο δύσκολες. Οπότε θα πρέπει να ε, φύγουμε από αυτό το ιστορικό μοντέλο των συνομότερων δυνατών και να πάμε σε ένα ενιαίο μοντέλο στρεματικής ενίσχυσης. Επίσης για τις ε, μειονεκτικές περιοχές. Στο Κοινοβούλιο πριν από ένα έτος εγκρίναμε μια έκθεση για τα προτινόμενα κριτήρια της Κομισιόν για τις μειονεκτικές περιοχές θεωρώ νομίζω πως ε, είναι σημαντικό και για τη δική σας τη χώρα αυτό το θέμα και έκτοτε υπάρχει νεκρική υγεία από την ε, Κομισιόν δεν έχουμε ακούσει τίποτα παρά το ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση εντός ενός έτους θεωρούν πως τα κριτήρια της Κομισιόν δεν είναι καθόλου καλά αντιθέτως είναι προβληματικά και φοβούμε πως ε, η όλη αυτή η υπόθεση βεβαίως θα χαθεί στην γενικότερη συζήτηση για την ΚΑΠ, αλλά το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω στην μεταρρύθμιση να δείτε αυτό το θέμα και εγώ απόρρισα για το ότι δεν υπήρχε ούτε λέξη στην ανακοίνωση Κομισιόν για αυτό το θέμα. Οπότε, από ό,τι φαίνεται θα περάσει έτσι σε σιωπή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Γιάρ και μετά ο κύριος Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σε εύχομαι καλή επιτυχία για τη μεγάλη ευθύνη που έχετε αναλάβει. Σε μια αποφασιστική φάση μιλάμε για τη μεταρρύθμιση θα έρθουν οι νομοθετικές προτάσεις. Μιλάμε ταυτόχρονα για τον προϋπολογισμό και νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό σε αυτή τη φάση μια νέα χώρα στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο η Γεωργία το ότι έχει αναλάβει την ε, Προεδρία. Και νομίζω πως ε, εσείς ε, είστε σύμμαχός μας στα ζητήματα της γεωργικής πολιτικής. Έχω δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη φορά τον προπολογισμό. Το πρώτο πρόβλημα που έχω νομίζω πως περνάμε σε μια παγίδα εδώ πέρα. Στην συζήτηση η Κομισιόν μιλάει για μια επιτυχία γιατί λέει πως κατάφερε να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός ε, της Γεωργίας αλλά βεβαίως οι γεωργοί μας αντιλαμβάνονται πως εγώ θα λαμβάνω ονομαστικά το ίδιο ποσό το 2013, αλλά είναι σαφές πως ε, μιλάμε για μία μείωση σε αυτή την περίπτωση κατά 14%. Οπότε, σας παρακαλώ να σπάσετε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για διατήρηση, να παραδεχτούμε πως πρόκειται περί μίας ε, μείωσης ή τουλάχιστον να το ξεκαθαρίσουμε πως μιλάμε ονομαστικά για το ίδιο ποσό γιατί βεβαίως ε, αλλιώς γινόμαστε αναξιόπιστοι. Εντάξει, και οι αγρότες ε, τα αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, για την ε, δικαιοσύνη όσον αφορά την κατανομή τα είπε και ο κύριος Ντόρφμαν, για εμένα η έκπληξη είναι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Εντάξει, το περίμενα, αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερε οι διαφορέ εντό ενό κράτου μέλους, κάτι το οποίο πραγματικά μου προξενεί έκπληξη. Και αυτό νομίζω είναι ζήτημα δικαιοσύνης ε, της ε, κατανομής για να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική, όχι μεταξύ κρατών μελών, αλλά και εντό των ε, κρατών μελών. Τελευταίο ερώτημα για τον προϋπολογισμό. Για τις άμεσες πληρωμές, τι άποψη για την ε, σταδιακή κατάργηση των άμεσων ε, πληρωμών κατόπιν για την ε, υγεία των ζώων και τη σήμαση των ζώων. Χάρηκα για το ότι αναφέρατε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να αναφέρουμε να δούμε αυτό το πρόβλημα, να υπάρξει λιγότερη γραφειοκρατία. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα είναι σήμανση στα πρόβατα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ε, πολλοί συνάδελφοι θεωρούν πως ε, υπερβάλαμε με τη γραφειοκρατία στα πρόβατα. Νομίζω θα πρέπει να ξαναδείτε το συγκεκριμένο θέμα γιατί εγώ θεωρώ πως ειδικά όσον αφορά την ε, σήμανση των προβάτων έχουμε επιβάλει μειονεκτήματα στις ε, μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Και ε, να συμφωνήσω με την κυρία Μαγκίνες στο θέμα των ε, συστοιχειών κλοβών των πουλερικών. Έχουμε πολύ διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλους στον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε γιαρο, ο κύριος Παπαστάνκος και κατόπιν ο Ιλίος Καπελσάντος. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και σας προσωπικά ε, καλή δύναμη κύριε Υπουργέ. Ε, το μήνυμα της χθεσινή μας συνάντησης με τον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Τσιόλος, το, αν μπορώ να συνοψίσω το μήνυμα της, ε, των συναδέλφων, ήταν ότι πρέπει να κινηθούμε ανωδικά σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 ε, σε σχέση με την πρόταση της, ε, της Κομισιόν. Ανωδικά και όχι καθοδικά. Ε, παρακολουθώ κύριε Υπουργέ τις ε, εξωτερικές πτυχές, τις εξωτερικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και επομένως και τις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Εμπορίου. Και επί της ουσίας προσυπογράφω όλα όσα είπε η καλή συνάδελφος η κυρία Μαγκίνες. Ε, για την ασφάλεια των προϊόντων, για την αμοιβαιότητα, για ισοδύναμους κανόνες. Αυτό θα πει δίκαιο εμπόριο. Ε, αυτό θα πει δίκαιη, ε, ισόρροπη διεθνής εμπορική τάξη. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα, οι οποίες έχουν κολλήσει και παρά την ε, άφθονη πολιτική δηλώσεων σε κάθε συνάντηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και στο G20 ότι ναι, όθηση, τίθενται χρονοδιαγράμματα, ε, δεν επαληθεύονται και ε, εκ νέου ανανεώσεις, συνεχείς ανανεώσεις προσδοκιών. Ε, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας και μαζί με τους συναδέλφους μια υπερκενοτόμο πρότασή μου, μια προθυμένη πρόταση. Ως γνωστόν, ο όγκος των ε, εμπορικών ροών των αγροτικών προϊόντων στην παγκόσμια κλίμακα είναι περίπου 7%. Αλλά είναι το πρόβλημα, είναι το αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για το γύρο της Δόχα, γιατί ως γνωστόν ο γεωρικός τομέας έχει ξεχωριστή σημασία για συγκεκριμένα κράτη, για συγκεκριμένες περιοχές, για συγκεκριμένα ε, προϊόντα. Και αυτό είναι κατανοητό όταν μιλούμε πολιτικά και συζητούμε, κάνουμε πολιτική ανάλυση. Η πρότασή μου η προωθημένη είναι, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι προεκτείνει το άλλο. Μήπως θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός διαπραγματεύσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, εκτός διαπραγματεύσεων του γύρου της Δόχα, το γεωργικό πακέτο και να προωθήσουμε τα υπόλοιπα όλα, όλα τα άλλα κεφάλαια από τη στιγμή που στόχος, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε, αφετηριακός στόχος των διαπραγματεύσεων του γύρου της Δόχα είναι η αρμονική ένταξη των απτυσσομένων χωρών στο διεθνές εμπόριο και μέσω αυτής της ένταξης η υποβοήθηση των απτυσσομένων χωρών. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ε, και πιστεύω ότι αν ολοκληρώσουμε τα άλλα κεφάλαια θα δοθεί και μια δυναμική στις διαπραγματεύσεις για το αγροτικό πακέτο. Και το δεύτερο είναι, μήπως πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε και η πρόταση πρέπει να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την καθίδρυση, τη δυνατότητα καθίδρυσης ενός παγκοσμίου ε, γεωργικού οργανισμού, ενός ξεχωριστού ε, δηλαδή, ε, οργανισμού γεωργίας, παγκοσμίου οργανισμού γεωργίας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και όσο αφορά τις προδιαγραφές ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων και βεβαίως και το εμπόριο αυτό καθευτό. Νομίζω ότι έτσι πως είναι τα πράγματα και η αρχιτεκτονική, η θεσμική αρχιτεκτονική, δηλαδή κάτω από την ομπρέλα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου πάρα πολλά θέματα, αδικούμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά δεν έχουμε και αποτελέσματα. Δηλαδή θα, θα μπορούσα να προσθέσω ότι σε αυτή τη λογική της παγκόσμιας, μιας νέας αρχιτεκτονικής, ότι χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό οργανισμό. Γιατί και το περιβάλλον, πολύ καλά προσπαθούμε και την οικολογική ευαισθησία και την ανάγκη οικολογικής πλαισίωσης και του εμπορίου ακόμα να την υπαγάγουμε, να την εντάξουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στην, ε, στην Προεδρία. Ευχαριστώ, κύριο Καπούλα Σάντο. Και κατόπιν ο αντιπρόεδρος Πουβέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ήδη είχα την ευκαιρία να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία, ιδιωτικά σε εσά, αλλά ήθελα να το κάνω και δημοσίω. Το Κοινοβούλιο <laughs> έχει μεγάλε προσδοκίε από την Πολωνική Προεδρία. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τι φιλοδοξίε που μας αποκαλύψατε και για το πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα της Προεδρία. και θα ήθελα να θέσω δύο σημαντικά ζητήματα θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η στρατηγική της Πολωνικής Προεδρίας ε, και το πρώτο το θέμα του προπολογισμού. Ξέρουμε ότι συμμερίζεστε τις ανησυχίες μας σε σχέση με την ανεπάρκεια της πρότασης της Κομισιόν σε σχέση με τον προπολογισμό της ΚΑΠ και θα ήθελα να μας πείτε ποιε πρωτοβουλίε θα αναλάβει η Πολωνική Προεδρία για να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη στην πρόταση αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τι είναι ισοτιμία. Είναι, ε, πρέπει να υπάρχει ισοτιμία σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις μεταξύ των κρατών μελών ή να προσπαθήσουμε τουλάχιστον προοδευτικά να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι είναι οι πρωτοβουλίες ε, σκοπεύει να αναλάβει η Προεδρία για να συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ Λουίς, ο κύριος Μποβέ και κατόπιν Νέιμερς. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τους επόμενους 6 μήνες ε, θα συνεργαστούμε με τον, Πολωνικό Υπουργό, με τον Πολωνό μας Υπουργό Γεωργίας και θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρος αυτή η συνεργασία γιατί όπως είπατε και εσείς η Πολωνία είναι μεγάλη γεωργική χώρα, έχει πάρα πολύ ε, ισχυρή αγροτική ιστορία και οι χωρικοί αγρότες ε, έχουν αγωνιστεί τα μάλα ε, για να πέσει ο κομμουνισμός στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν πρέπει να χαιρετήσουμε το σημαντικό αυτό πολωνικό κίνημα, του Solidarnosc. Θα ήθελα να επιμείνω σε μια σειρά σημείων το θέμα της ε, ισότητας ε, στην ε, κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των διάφορων κρατών μελών. Αναφέρθηκε από πολλούς και νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να έχουμε αυτή την ισοτιμία μεταξύ των χωρών και των γεωργών για να έχουμε μια γεωργική Ευρώπη. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε και από τον Επιτροπό Τσόλος. Νομίζω ότι αυτή συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων από τη δική σας Προεδρία και στο βαθμό που η Πολωνία έχει μεγάλο αγροτικό ιστό, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα είναι πολύ σημαντικό και για σας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο ζήτημα που θέλω να προσεγγίσω έχει να κάνει με το θέμα της βιομηχανικής γεωργίας, γιατί και εσείς ε, συνδέσατε το θέμα αυτό με το περιβάλλον και με τις διεθνείς αγορές. Σήμερα ανησυχούμε για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλες, ε, όμιλοι, με συγχωρείτε, Σμίθφιλ, παραδείγματος χάρη, ε, ουσιαστικά πώς ε, επί ε, συγκεντρώνουν την αγροτική παραγωγή και τη ζωική παραγωγή και συγκεκριμένα αναφέρουμε ε, στο χοιρινό κρέας και συμβαίνει και στην Ανατολή και στην Πολωνία και στην Ρουμανία αλλά και σε άλλες χώρες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι διεξάγουν κάποιες πολιτικές που είναι αντίθετοι στα συμφέροντα των οργανώσεων των αγροτών. Τρίτο θέμα, ε, και σας το θέμα, αλλά όχι σε βάθος. Ε, θα συζητήσουμε και πάλι για τους γενετικά τροπομένους οργανισμούς. Ε, ξέρετε, συγγνώμη, για για του ε, γενετικά τροπημένου οργανισμού, λοιπόν, το συστήσαμε και εμεί την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα, λοιπόν, να, να μου πείτε και ποια είναι η δική σα γνώμη σχετικά με την απαγόρευση των γενετικά τροπομένων οργανισμών. Ευχαριστώ, Ζωζέ, Ρέιμερ και Όσλινγκ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, για να έχουμε μαζί την ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να αναφέρθω και εγώ σε κάποια πράγματα που ήδη ακούστηκαν από τη μία λέμε το ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη γεωργία στις ε, εμπορικές συναλλαγές, αλλά από την άλλη η κυρία Μαγκίνε, σωστά ανέφερα πως ε, πρέπει να δούμε την ε, ενιαία εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι πράγματι η κλοπή των πουλερικών και νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό και για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, προς τα έξω. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν ζητάμε προδιαγραφές και τήρησή τους ε, όταν δεν είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε εντός της Ευρώπης. Υπάρχει εδώ πέρα ανάγκη να γίνει πρόοδος, σημαντική πρόοδος. Και θα πρέπει να εκπληρώσουμε αυτές τις ε, προδιαγραφές. Το δεύτερο χαιρετίζω βεβαίως το πόσο σημαντική είναι για εσάς η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων γιατί νομίζω πως ε, στο μέλλον θα ε, έχει μεγαλύτερη σημασία η ασφάλεια των τροφίμων. Είναι σαφές πως αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός και άρα η ανάγκη για τρόφιμα και στην Ευρώπη νομίζω πως είμαστε σε καλή θέση για παραγωγή τροφίμων και δεν πρέπει να το παραμελήσουμε αυτό, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Κατόπιν, να υπενθυμίσω πως όταν μιλάμε για τη δίκαιη κατανομή μέσων, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ε, σταδιακή μείωση των ε, πληρωμών, γιατί βέβαια υπάρχει και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Να υπάρχει δηλαδή μια κλιμάκωση. Γιατί επίσης Ε, να δούμε και το ζήτημα των ε, καυσίμων γιατί εάν ε, δεν λυθεί αυτό το ζήτημα όπως επίσης και το ζήτημα των μειονεκτικών περιοχών θα δημιουργηθούν πολλές δυσαρέσκειες γιατί δεν είναι πάντα αυτό το οποίο εμείς προφανές, προφανώς θεωρούμε μειονεκτική περιοχή όντως μειονεκτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρτίν Όσλινγκ και κατόπιν Αλμπερτές. Ναι, κύριε Υπουργέ, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τώρα το ερώτημα. Το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ της μεταρρυθμίσης γεωργίας. Πόσο γρήγορα εκτιμάτε πως ε, θα καταλήξει μια ανάλογη θέση και το Συμβούλιο, γιατί ο χρόνος πιέζει. Και Το ερώτημα είναι πώς θα ακολουθήσετε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και να βρείτε κάποια συμφωνία με το Συμβούλιο. Το ερώτημα πολλών είναι βεβαίως ε, το ζήτημα ενός ε, κάποιων ε, περικοπών ή ενός ε, πλαφών. Ε, θα δούμε τι θα γίνει. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η στάση τη σας γιατί υπάρχει βέβαια και το θέμα των θέσεων εργασίας. Κατόπιν αναφέρατε το θέμα των σπόρων και το τι θα έρθει τώρα από την Γενική Διευθυνσή ΣΑΝΚΟ. Υπάρχει κάποια πρόταση. Πρέπει, λέτε, να υπάρξει κάποια απελευθέρωση στην Ευρώπη και να γίνουν τα πράγματα απλούστερα τι απόψεις έχετε. Δεν σας κρύβω πως ε, μας ανησυχούν κάψως οι απόψεις της ε, Κομισιόν. Την δε προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την μελλοντική πολιτική όσον αφορά τα ε, γεννητικά τροποιημένα τρόφιμα και την έκθεση Λεπάζ. και για την προστασία της ε, γεωργίας ελεύθερης από γενικά ε, τροποποιημένους οργανισμούς. Και τέλος το είπε και η κυρία Ρόντου στο θέμα του γάλακτος. Από τις δηλώσεις σας καταλαβαίνω πως δεν είστε ικανοποιημένος με το status quo και από ό,τι φαίνεται δεν είστε ικανοποιημένο όσον αφορά αυτή την ε, ήπια προσαρμογή. Τι απόψε έχετε για τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για το χρόνο μετά το 2015. Ο και μετά ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το ότι απουσίαζα, αλλά προσπάθησα να έρθω ξανά. Από το 1990, κύριε Υπουργέ, ως Γερμανός βουλευτής τότε είχα επισκεφτεί πολλές φορές ε, τη χώρα σας και από το 2004 ως Ευρωβουλευτής και πάντα μου προξενεί έκπληξη η θετική ανάπτυξη της χώρας σας. Ήμουν πάντα στην Ήπεθρο και σε κάθε επίσκεψη μετά από ένα ή δύο χρόνια βλέπαμε πραγματικά την εξέλιξη της Πολωνίας με τι όρεξη προσπαθούσαν ειδικά οι νέοι να προοδεύσει η Πολωνία. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό κύριε Υπουργέ τώρα που έχετε την ε, Προεδρία θα φροντίσετε την κοινή γεωργική πολιτική και για εμένα αντιπροσωπεύετε την ελπίδα για το ότι η γεωργική πολιτική θα προοδεύσει αυτό το εξάμεινο και στο τέλος θα έχουμε ένα αποτέλεσμα και με εντυπωσίασε αυτό το οποίο είπατε, πως δεν είναι δυνατόν στο τέλος αυτών των ε, διαπραγματεύσεων να έχουμε πάλι περισσότερη γραφειοκρατία για τους ε, αγρότες και θα πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε άρα προς αυτή την κατεύθυνση της απλούστερης γεωργικής πολιτικής. και θέλω να το ξαναπώ και σήμερα δημοσίως πως χρειαζόμαστε μια ισχυρή ε, γεωργία για να θρέψει το μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους, ε, να παράγει ανανεώσιμες φυγές ενέργειας και βεβαίως ένα πράγμα πρέπει να τονίσουμε και χαίρομαι που το είπατε σήμερα πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στην κοινή γνώμη πως η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι παγκοσμίω η πιο αηφόρος που υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που πρέπει να καταπολεμήσουμε και νομίζω πως θα έχουμε τις επόμενες 6 μήνες μια καλή ε, συνεισφορά από το πλευρό σας και νομίζω πως ε, το ΕΛΚ θα συνεργαστεί με τους ε, Πολωνούς συναδέλφους να σας στηρίξει. Ευχαριστώ, Άλμπερτ, ο κύριο Νίκολσον. Και μετά, κύριε Γιώσο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο θα αναφερθώ σε ορισμένα θέματα. Καταρχήν, Καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή καθώς ε, ανακοινώθηκαν τώρα οι δημοσιονομικές προοπτικές όταν ε, εγώ εκλεκτικά σε αυτό το κοινοβούλιο, η ΚΑΠ ήταν άνω του 65% του προπολογισμού, σήμερα είναι 39, κάτι του προπολογισμού. Πού βλέπετε να βρίσκεται το 2020? Δηλαδή, αν ε, συνεχιστούν ε, τα πράγματα στις MPS ε, όπως ήταν τα τελευταία 20 χρόνια, τι θα γίνει με την ασφάλεια, την επιστηστική σε 10 χρόνια. Αυτή είναι η ερώτηση στο μυαλό όλων, γιατί η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι αν δεν υποστηρίξετε την παραγωγή τροφίμων μέσω της αρρωγής στο Γιώργο, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω στα σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε και αν αγοράζει τα τρόφιμα αυτά, γιατί δεν δεν υπάρχουν φτηνά τρόφιμα και θα πρέπει να πληρώνουμε για αυτά τα τρόφιμα. Επίσης να προσθέσω τη φωνή μου σε όσους είπαν ε, ότι Ε, θα έχετε, παραδείγματο για αυτή την ε, απαγόρευση, ε, θα πρέπει να εργαστείτε για να μπει σε εφαρμογή από του χρόνου τον Ιανουάριο και αν τελικά δεν διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει εφαρμογή, τότε θα δώσουμε πολύ κακή εντύπωση. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το πακέτο για το γάλα γιατί εγώ ήμουν υπεύθυνο, είμαι υπεύθυνο για το το γάλα και έχουμε τώρα μια γενική εικόνα για το που βρισκόμαστε, όμως το πακέτο αυτό έχει να κάνει με τους παραγωγούς και έχει να κάνει και με τους μεταπίτες, με τους επεξεργαστές, θα πρέπει αυτοί να συνεργαστούν. Το μόνο που δεν καλύπτει και εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό ε, και είναι ο γενικός τομέας. Έτσι λοιπόν τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να επανέλθει και να μου πει ε, ότι θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα το 2017 γιατί θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή για δύο χρόνια και θα χρειαστει δωδεκάμενη αξιολόγηση για το πώς θα λειτουργεί η νομοθετική πρόταση. Αλλά φοβάμαι ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό ότι δεν θα μπορέσουμε να ελέγχουμε ε, την κατάσταση στην αγορά. Θα έχουμε έκρηξη στην αγορά του γάλακτος και πώς θα είναι η κατάσταση και πώς θα το ελέγξουμε αυτό. Γιατί αυτό είναι ο μεγάλος μου φόβος σε σχέση με το τι κάνουμε. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπε, είπε η Μαριάν Σίφερμπολ για την ομαλή προσγείωση για το γαλακτοκομικό τομέα. Και όταν μιλώ σε κάποιους θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν ε, αυτή την ομαλή προσγείωση και θεωρούν ότι ούτε καν κοντά είμαστε σε κάτι τέτοιο. Ε, θα πρέπει να συνεργαστώ μαζί σας ε, και με το Συμβούλιο για να το πετύχουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό το πακέτο για το γάλα. Γιατί αν περάσουμε στις συμβάσεις από τις ποσοστώσεις θα πρέπει να βρούμε μία λύση που να λειτουργεί και για τους γεωργούς. Ευχαριστώ Τζιμ. Κυρία Γιούζα και κατόπιν Ολενίτσικα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία γιατί έχετε δύσκολο έργο μπροστά σας. Εγώ συμφωνώ μας είπε η κυρία Μαγκίνες και θα ήθελα να κάνω κάποιε σκέψει. Ε, ο προπολογισμό της κοινή αγροτική πολιτική στην καλύτερη περίπτωση θα διατηρηθεί παγωμένο με ένα προπολογισμό που έχει προβλεφθεί για κάποιε χώρε. Όμω ε, η προοπτική δεν είναι καλή για του αγρότε. Κάθε φορά είναι μικρότερο το εισόδημα και οι γεωργοί πρέπει να πληρώνουν όλο ένα και περισσότερο για τις ζωοτροφές, τα φυτοφάρμακα, έχουν υπερβολικό κόστος παραγωγής, αν συγκρίνουμε τι συμβαίνει με τις ανταγωνιστικές ε, χώρες. Απλώς ε, επειδή εμείς έχουμε αυστηρή νομοθεσία για την ευημερία των ζώων, ε, όλης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της απαγόρευσης των γενικά τροπημένων οργανισμών. Επίσης έχουμε στην Ευρώπη το πρόβλημα της τροφικής αλυσίδας η συγκέντρωση της διανομής είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά των τιμών ε, μεταξύ το τι εισπράττει ο αγρότης και το τι πληρώνει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ είναι τεράστια. Εγώ δεν ε, ξέρω πώς ε, η δική σας προεδρία θα το προσεγγίσει το θέμα αυτό. Επίσης, ακούστηκαν πολλές παρεμβάσεις σε σχέση με τις διαφορές κατανομής, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στο εσωτερικό μιας χώρας. Η Προεδρία σας πώς θα το προσεγγίσει το πρόβλημα αυτό, θα λάβετε υπόψη τις αντίξωες συνθήκες ορισμένων περιοχών, γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο εγκατάλειψης Δηλαδή η Γεωργία όχι μόνο δεν θα είναι, αποφέρει πλέον έσοδα, αλλά θα, θα υπάρχει και ελάχιστο εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει κάποιο από τη Γεωργία. για μιλήσατε ε, για τα τρόφιμα. Δεν πιστεύετε ότι πέρα από την ε, πρόθεση που κάνουμε σε τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνει και πρόθεση έτσι ώστε η κατανάλωση ευρωπαϊκών προϊόντων να γίνεται και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί στην Πολωνία είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που δεν γνωρίζουμε στην Νότια Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι η αυτοκατανάλωση δηλαδή των ευρωπαϊκών προϊόντων θα είναι πολύ σημαντική για την ε, πρόθεση των τροφίμων και επίσης αν πουλάμε τα αγαθά μας μέσα στην Ευρώπη, αντί να εξάγουμε σε τρίτες χώρες, θα μειώσουμε και τις εκπομπές. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, εγώ περιμένω τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγιούζο. ο κύριος Ολένιτσεκ και μετά ο George Λάιον, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Υπουργό. Λυπάμαι που δεν ε, ήμουν νωρίτερα στη συνεδρίαση γιατί Ήμουν στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου ακούσαμε την αρμόδια Πολωνέζα Υπουργό εκεί. Θα ήθελα να σας συγχαρώ πάντως ε, για τη στάση που κρατάτε και για την ε, δέσμευσή σας να προωθήσετε θέματα που και για μας ε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, στην Επιτροπή Γεωργίας δηλαδή και το πακέτο που μας παρουσιάσατε ανταποκρίνεται πλήρως και στις ανάγκες και ενδιαφέροντα της δικής μας Επιτροπής. Νομίζω ότι έχουμε όλοι μεγάλη τύχη που στη διάρκεια τη της κρίσης και σε δύσκολη στιγμή των διαπραγματεύσεων για γεωργική πολιτική αναλαμβάνει την Προεδρία, η Πολωνία και μάλιστα εσείς συγκεκριμένα κύριε Ζαβίσκη γιατί η θέση και η δική σας και του Υπουργείου σας είναι γνωστή και εκτιμάται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι μπορούμε να ανακεφαλώσουμε τη θέση μας στο ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα για την κοινή γεωρική πολιτική και την ε, καλύτερη κατανομή αυτών των κονδυλίων ε, ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους ε, κλάδους της γεωργίας ώστε να αναπτυχθεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Έτσι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη θέση σας. Επίσης ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί έχουμε ε, και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το πολύ καλό επιτελείο που έχουμε στη διάρκεια, θα έχουμε στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, γιατί και το προσωπικό σας επιτελείο, οι συνεργάτες σας είναι πολύ αξιόλογοι και εσείς θα τους οδηγήσετε με πολύ στιβαρό χέρι. Και θα ήθελα να εκφράσω την ευχή μου το δυναμικό αυτό να αξιοποιηθεί και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πακέτο Θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομοθετικό πακέτο ώστε να το αναλάβει το συντομότερο δυνατό η Πολωνική Προεδρία. Γιατί οι πολωνικέ προτεραιότητε, οι προτεραιότητε τη Πολωνική Προεδρία ε, αναφέρονται στο νομοθετικό πρόγραμμα. Αν δεν υποβληθεί αυτό το νομοθετικό πακέτο, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα, ούτε θα μάθουμε τη θέση των υπόλοιπων χωρών μελών σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία αυτού του νομοθετικού πακέτου. Πρέπει να πρώτα το πακέτο λοιπόν. Από αυτή την άποψη υπάρχουν ελπίδες να υποβληθεί το Σεπτέμβρη, το αργότερο τον Οκτώβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το νομοθετικό πακέτο. Ποιες είναι οι δικές σας προβλέψεις σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε και χθε τη θέση της για τον γεωργικό προϋπολογισμό. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Θα γίνει πεδίο μάχης ε, ε, θα γίνουν πεδίο μάχης ε, αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θα υποστηρίξετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γεωργικό προϋπολογισμό. Γιατί τη δική σας θέση την ξέρουμε. Ε, βέβαια, σας περιμένατε ακόμη μεγαλύτερο κονδύλιο για τη γεωργική πολιτική και δικαίως, αλλά ε, ποια είναι η θέση και των υπόλοιπων κρατών μέλων και ποια θέση θα κρατήσετε εσείς στο Συμβούλιο. Επίσης, υπευλήσαν ερωτήσεις για το πακέτο ποιότητας των τροφίμων. Πότε θα αναλυθούν δράσεις και στον τομέα αυτό. Και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό της προτάσεις της για την προαγωγή, την προώθηση. Γιατί η Πολωνία έχει πολύ πλούσια πείρα που θα μπορούσε να την, ε, να την αξιοποιήσουν και οι υπόλοιπε χώρες. Γιατί προωθούμε και διαφημίζουμε πολύ καλά τα προϊόντα μας και τα διαθέτουμε και σε άλλες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διδαχθεί από τις δικές μας θετικές εμπειρίες. Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ επίκαιρο και ε, ενδιαφέρει φυσικά και την Πολωνική Προεδρία. Θα πρέπει να γίνει κάτι και στη σχέση μας με τη Ρωσία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις πωλήσει. Απευθύνω έκκληση σε όλες τις χώρες μέλη και στους ευρωβουλευτές να επιδείξουν αλληλεγγύη γιατί αυτή τη στιγμή μόνο μερικές χώρες μπορούν να διαθέσουν νοπά απορροκυπευτικά για να πουλήσουν προς τη Ρωσία ενώ άλλες χώρες δεν δίνανται να πουλήσουν νοπά απορροκυπευτικά προς τη Ρωσία. Πώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις κύριε Υπουργέ με τη Ρωσία. Έθεσε ορισμένε ερωτήσει, έκανα κάποιε παρατηρήσει. ήθελα και πάλι να σα συγχαρώ και να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση, γιατί σε αυτή την αντίξωη και δύσκολη στιγμή έχουμε την τύχη να ε, συμμετέχουμε στην Πολωνική Προεδρία, να γινόμαστε μάρτυρε της Πολωνικής Προεδρίας και να σας συγχαρώ θερμά και σα προσωπικά αλλά και το πολύ αξιόλογο επιτελείο σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε George Lyon. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μια απάντηση για τον προτεραιόμενο προπολογισμό από την Κομισιόν και αυτή τη νέα δομή όπου έχουμε σχεδόν 15 δισεκατομμυρία λίρες ε, που θα βγουν ε, από τη συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού στην πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ αυτά τα χρήματα για αγροτικούς σκοπούς και αν θα ωφεληθούν οι γεωργοί. Αναρωτιέμαι ποια είναι η αντίδρασή σας ε, σε αυτό το τρίτο αποκαλούμενο πυλώνα του προπολογισμού φαίνεται να εισαγάγεται τώρα μέσω των προτάσεων ε, της Κομισιόν. Γιατί σίγουρα δεν έχουμε σαφή ένδειξη για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Πιέσαμε τον Επίτροπο χθε για το θέμα αυτό και του είπαμε τι θα γίνει με τα χρήματα αν δεν δαπανηθούν ε, στο οικονομικό έτος, ε, θα εξαφανιστούν αυτόματα σε άλλους τομείς του προπολογισμού. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω για την πρόταση της Κομισιόν είναι μία πρόταση να αναλαμβάνουν τις αποφάσεις τα κράτη-μέλη σε σχέση με την καλλιέργεια μικρών. Το Κοινοβούλιο κατέληξε τελικά, κατέκπληξε στην υποστήριξη αυτή της ιδέας. Πώς σκοπεύετε εσείς να προχωρήσετε στο θέμα αυτό. Και αν να μας πείτε αν θα είναι προτεραιότητά σας να σημειώσετε πρόοδο στο θέμα αυτό μαζί με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Τζόρτς. Αγαπητέ Πρόεδρε, ακούσατε τις ε, παρεμβάσεις. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλά λεπτά θέματα, αλλά και φιλοδοξίες αυτής της Επιτροπής επίσης είναι πολλές. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε το επόμενο εξάμεινο της Πολωνικής Προεδρίας να μπορέσετε πράγματι να καταλήξετε σε σημαντικά αποτελέσματα. Έχετε το λόγο για τις απαντήσεις. Panie Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να πω ότι άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Άκουσα τις απόψεις σας και ως Γιώργος ε, και Ευρωβουλευτής ε, και Βουλευτής, συγγνώμη, πάρα πολλά χρόνια έχω ε, την πεποίθηση ότι υπάρχει ευκαιρία και υπάρχει πρόσφορο έδαφος ε, για ευόδοση των ε, συζητήσεων για την κοινή γεωργική πολιτική. Για τη συζήτηση αυτή βέβαια θα πρέπει να βρούμε χρόνο και θα πρέπει από κοινού να, να δείξουμε και η όβια υπομονή. Σήμερα βέβαια συμμετέχω εδώ ως προεδρεύων του Γεωργικού Συμβουλίου. Συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας και δεν μπορώ να ε, εκφράσω ιδιαίτερα προσωπικές αποφάσεις. Βέβαια, πολλοί με ρώτησαν και για τις προσωπικές μου θέσεις, γι' αυτό και δεν μπορώ να το αγνοήσω. Πάντως, ο ρόλος μου είναι, όπως είπα και στην αρχή, πρώτον, να εξασφαλίσω καλές συνθήκες συνεργασίας για επίτευξη συμβαστικής λύσης ε, στο Συμβούλιο, αλλά πρώτα απ' όλα, και μην προσβληθείτε από αυτό, την εκμετάλλευση της αξιοποίησης ε, της ε, διάθεσης και του δυναμικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ιδιαίτερα της Επιτροπής Γεωργίας, ώστε ως ισότιμοι εταίροι να συνεργαστούμε και να λάβουμε από κοινού αποφάσεις που θα είναι θετικές για τη γεωργία, τους γεωργούς, αλλά και για τους καταναλωτές. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι εμείς οι γεωργοί δεν παράγουμε για τους εαυτούς μας, δεν εργαζόμαστε μόνο για την προσωπική μας ικανοποίηση, πρώτα απ' όλα εργαζόμαστε για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές είναι σημαντικότεροι για μας και σε αυτούς απευθύνεται το έργο και η δουλειά μας. Οπότε σιγά σιγά θα έλθω στις ερωτήσεις που θέσατε και όπως είπε και ο Πρόεδρος στην αρχή, ξεκινάμε τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής σε όρους και συνθήκες που καθορίζονται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προτάσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς ε, έχουμε καθυστερήσει τουλάχιστον μια διετία σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την κοινή πολιτική. Γιατί το 2008 είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία για μια επισκόπηση της κοινή γεωρικής πολιτικής ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη διετία που πέρασε και να διευκρινίσουμε ακριβώς τι θέλουμε να αλλάξουμε με τη μεταρρύθμιση αυτή. Αλλά περιμέναμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Χάσαμε αυτή τη διετία και σήμερα έχω σοβαρές ανησυχίες ότι όλοι όσοι ε, καθόμαστε εδώ και βρισκόμαστε εδώ θα γίνουμε όμοιροι τη συζήτηση του δημοσιονομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει κάπως να τα συνδυάσουμε και να τα συμβάσουμε. Θα πρέπει να βρούμε συμβαστικέ λύσεις για τη γεωργία στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι και μόνο το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει προτάσει που ικανοποιούν ε, την βασική προτεραιότητα της κοινή πολιτικής που είναι η απλούστευσή της. Γιατί από δύο πυλώνες ε, που είχαμε μέχρι στιγμής εμείς είπαμε ότι δημιουργείται και κάτι τρίτο, ένα τρίτο, ένας τρίτος πυλώνας, αυτό που θα απομείνει υποτίθεται υπό την ε, επιρροή της Γεωργίας και της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, αλλά στην ουσία έχει προκύψει από κάπου πιο μακριά. Δεν θα αποφασίσει η Γενική Διεύθυνση Αγκρή για το πώς ε, αυτά τα αποσυνδεδεμένα δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν. Μερικοί από εσά ε, ανέφεραν αυτούς τους φόβους και ο George Lyon το έκανε. Ε, λοιπόν και εκφράσαμε τους φόβους αν αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στους Γεωργούς γιατί ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι κατευθυντήριες αυτές τις προτάσεις του δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι και για μας θετικές. Ο κύριος, ο κύριος Παπαστάμκος ο κύριος Παπαστάμκος λοιπόν αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και στην εξωτερική πολιτική, στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα, στις διαπραγματεύσεις για το Μερκοσούρ. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι σήμερα η Γεωργία είναι στην ουσία αντικείμενο στην αγορά του εμπορίου. Σήμερα η Γεωργία αντιμετωπίζεται ως όμοιρος, ως εχμάλωτος στη συζήτηση των υπηρεσιών και σε θέματα που δεν έχουν σχέση με τη γεωργία. Και πραγματικά δεν φανταστώ ότι μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη γεωργία από αυτή τη συζήτηση. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει όμοιρος η γεωργία, να γίνει εχμάλωτος στους δύο αυτούς τομείς. Και πολύ εκφράσατε τον προβληματισμό και την ανησυχία σας για θέματα ασφάλειας, ποιότητας, τις απαιτήσει που επιβάλλουμε στους ε, Ευρωπαίους γεωργούς και αναφερθήκατε στην απελευθέρωση και στο άνοιγμα του εμπορίου προς προϊόντα για τα οποία δεν ισχύουν αντίστοιχες απαιτήσει. Πρόκειται για παραγωγές ε, που πολύ συχνά γίνονται υποσυνθήκες που καταστρέφουν το περιβάλλον, ενώ εμείς το φροντίζουμε και το προστατεύουμε στην Ευρώπη, και αναφέρθηκε και το θέμα για των εργασιακών συνθήκων. Οι τέτοιου είδου μερικέ φορέ εξοκοινωτικέ παραγωγέ δεν τηρούν καν τι στοιχειώδει συνθήκε του εργατικού δικαίου. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πολύ εντελεχή συζητήσει. Αν είναι τόσο υψηλέ οι απαιτήσει που επιβάλλουμε στου Ευρωπαίου γεωργού, τότε δεν θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχε απαιτήσει και υψηλέ προδιαγραφέ και για τα προϊόντα που εισάγουμε, για τα εξωκινοτικά προϊόντα. Τότε πραγματικά και οι δικοί μα γεωργοί θα έρθουν σε ίσου όρου με του εξωκοινωτικού παραγωγού. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στρατηγική, στρατηγική για τον προπολογισμό. Σίγουρα η συζήτηση μόλις τώρα ξεκινάει και κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει προδιαγραφεί, δεν έχει προεξοφληθεί. Βέβαια, σίγουρα από εμά, όλου εδώ, αλλά και από το Συμβούλιο, θα εξαρτηθεί αν θα καταφέρουμε να πείσουμε του οικονομολόγου, του πολιτικού, του φορολογούμενου, αν θα καταφέρουμε να του πείσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική αξίζει έναν προϋπολογισμό, θα είναι τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο και αν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε και να κατανείμουμε ορθολογικά αυτόν τον προϋπολογισμό. Τώρα, αν με ρωτάτε για την προσωπική μου γνώμη και τις θέσεις μου για τις άμεσες ενισχύσεις, γιατί πολλοί το ρώτησαν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Σε μια κατάσταση όπου η γεωργή της Λετωνίας λαμβάνουν 90 ευρώ ανά εκτάριο. Οι, οι Γάλλοι 350 ευρώ το εκτάριο και οι Έλληνες 560 ε, ευρώ το εκτάριο. Ερωτώ λοιπόν, αυτή η πολιτική είναι δική Και αν μετά την ε, αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή. Για παράδειγμα, ο τομέας ε, του χείριου κράτους που έχει έλλειμμα και οι, περισσότεροι, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη ευτυχώς βιομηχανική παραγωγή, αλλά έχουν ε, μικρές ε, εκμεταλλεύσεις. Υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες ανταγωνισμού σε μια ενιαία αγορά που η τιμή θα είναι ενιαία και με συνθήκες όπου οι πληρωμές ε, σε προϊόντα κρυθάρια, παράδειγμα, σε δημητριακά, είναι τριπλάσιες από ό,τι στην Λετωνία. Είναι δυνατόν να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό με τέτοιες συνθήκες στην αγορά. Επίσης, η κοινή γεωρική πολιτική με τη σημερινή της μορφή, στη σημερινή της εκδοχή. Δεν ήταν πολύ κλειστή και εγκλωβισμένη σε ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο. Και τελικά η κοινή γεωρική πολιτική είναι μόνο κατόνομα σήμερα η γεωρική πολιτική. Ε, Αναφέρθηκε το θέμα της ε, εξίσωσης των ε, ενισχύσεων στις διάφορες περιοχές και μεταξύ των διαφόρων χωρών. Είναι αλήθεια. Είπα πολλές φορές ότι σήμερα δεν έχουμε κοινή γεωργική πολιτική, δεν έχουμε ουσιαστικά κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε μόνο κατόνομα μια κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί στην ουσία δεν έχουμε 27 διαφορετικές γεωργικές πολιτικές, αλλά δεκάδες διαφορετικές γεωργικές πολιτικές. Και δεν μπορούμε καν να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Είναι τόσες πολλές και διαφοροποιημένες που δεν μπορούμε καν να τις συγκρίνουμε. Και αν σήμερα αναζητήσουμε πηγές ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία, εγώ επαναλαμβάνω ότι η γεωργία μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη γεωργία με, και με βραχυπρόθεσμη προοπτική δηλαδή ε, με το 2020 και με μακροπρόθεσμα το 2050. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τη συνήθεια της διαμόρφωσης ε, των ε, ενισχύσεων με βάση τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην πρώτη φάση της κοινή γεωρικής πολιτικής, το, θέμα, το θεμελιώδες θέμα ήταν η αύξηση της παραγωγής και η εξασφάλιση του επιστηστικού ανεφοδιασμού, γιατί τότε είχαμε έλλειμμα τροφίμων, ενώ τις τελευταίες ε, τα τελευταία 20 χρόνια δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τα πλεονάσματα και δεν μπορέσαμε να τα διαθέσουμε κατάλληλα στην ευρωπαϊκή αγορά. Είχαμε αντίθετο πρόβλημα. Και σήμερα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο και τελείως διαφορετικές ανάγκες. Σχεδόν όλοι και από παντού μας λένε ότι το 2050 θα χρειαστούμε κατά 80 ή 100% περισσότερα τρόφιμα από σήμερα. Τι σημαίνει αυτό. Από κάπου θα πρέπει να τη τα βρούμε αυτά τα τρόφιμα, κάπου θα πρέπει να τα παραγάγουμε αυτά τα τρόφιμα. Οπότε, ε, με απερίμωση των δασών ή με εξορθολογισμό της γεωργίας στις περιοχές που σήμερα υπάρχει γεωργική παραγωγή, κάνοντας μία αξιολόγηση, μία αξιολόγηση του δυναμικού της πιθανής αύξησης της παραγωγής και εντός της Ευρώπης. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε περιοχές που έχουν δυσμενείς συνθήκες για τη γεωργία. Αυτό ο μηχανισμός που εμπίπτει σήμερα στο δεύτερο πυλώνα λειτουργεί. Ανέφερα επανειλημμένως ότι οι ενισχύσεις για ε, περιοχές με αντίξωες συνθήκες και στηρίζοντας μία ισορροπημένη ακυφόρο γεωργία και δίνοντας ευκαιρία στη γεωργία και στις ε, ε, πιο δύσκολες περιοχές, δημιουργεί ε, ευκαιρία σε συγκεκριμένους γεωργούς συγκεκριμένων περιοχών να αναπτύξουν γεωργική δραστηριότητα. Και αυτές οι ενισχύσεις, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ανήκουν στον πρώτο πυλώνα και στις άμεσες ενισχύσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη για τις άμεσες πληρωμές, άμεσες ενισχύσεις, θα ήθελα να σας πω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεμβρίου αναφέρεται το, ο, το θεμελιώδες, ο θεμελιώδης συντελεστής. Εγώ λέω ότι το θεμελιώδης στατικό είναι η επιφάνεια της αρατρέας καλλιέργειας. Και Δύο ε, είναι ο συντελεστής και επίσης θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και τις συνθήκες ε, της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ε, των περιφερειών και να λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον, αν θέλουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε τη γεωργία και για τις επόμενες γενιές, ώστε να έχουμε ε, περιορισμού παραγωγών σε ορισμένες ε, γεωργικές ζώνες κοντά σε ε, προστατευμένες περιοχές και την τιμή, τη, τα σπασμένα μην τα πληρώνει συγκεκριμένη γεωργία. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δείξουμε το θάρρος και να θεσπίσουμε νέο σύστημα μέσω ενισχύσεων που θα στηρίζεται σε τέτοιο σύστημα, σε πιο αντικειμενικά κριτήρια. Και αυτό το συζητούμε στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα, γιατί στον πρώτο πυλώνα βρίσκονται τα περισσότερα κονδύλια. Γιατί όλη αυτή τη μάχη δίνουμε για όσο το δυνατό περισσότερα κονδύλια στη Γεωργία. Κατά τη γνώμη μου, στα πλαίσια αυτού του πρώτου πυλώνα και με βάση το σχέδιο που σας υπέβαλα, θα μπορούσαμε να πληρώνουμε στους γεωργούς για τις υπερβολικές ε, προδιαγραφές που τους απαιτούμε για την ποιότητα των τροφίμων, την, ε, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων, γιατί αυτά ε, μπορούν να καταμετρηθούν και για συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά και για συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα κονδύλια στην καινοτομία, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στην ανταγωνιστικότητα, στις νέες προκλήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτές οι προαιρετικές ε, δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται στο δεύτερο πυλώνα. Είπε κάποιο ότι 90% των κονδυλίων ε, βρίσκονται στον πρώτο πυλώνα. Έχω την αίσθηση ότι όλοι οι γεωργοί ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, όταν πριν από λίγο κυρία Ντές μιλήσατε για την επιτυχία της Πολωνίας, της πολωνικής υπαίθρου και των πολωνών γεωργών. Ε, ένας από τους λόγους της επιτυχίας ήταν το γεγονός ότι χάρη στον ε, ε, Ευρωβουλευτή Καλινόφσκη που ήταν ο διαπραγματευτής για τη Γεωργία στην Πολωνία, υιοθετήσαμε ένα σύστημα όπου τα μισά κονδύλια δίνονται σε πραγματικά ενεργούς γεωργούς. Και ενεργός γεωργός δεν είναι αυτός που παράγει μόνο για την αγορά ενώ μη ενεργός ε, γεωργός είναι αυτός που έχει ε, μόνο υπόψη την καινοτομία. Εμείς στα, προ... στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου δώσαμε ε, δυνατότητες στους γεωργούς 40% οι πιο ηλικιωμένοι, 60% οι πιο νέοι ενισχύσεις για εξυγχρονισμό, για επενδύσεις στις γεωρικές τους εκμεταλλεύσεις. Γι' αυτό η πολωνική ύπεθρος άλλαξε τόσο δραστικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι από αυτή την εμπειρία που είχαμε, αυτή την εμπειρία που είχαμε τη θετική θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε και στην Ευρώπη και να την αξιοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά την ακριβωδική κατανομή των κονδυλίων. Κατά τη γνώμη μου, η δίκη καταβολή δεν θα γίνει με βάση την εξίσωση, γιατί άλλοι λένε 90 χωρίς ανώτατο όριο. Ε, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος, αλλά θα πρέπει να βρούμε νέα αντικειμενικά κριτήρια. Ίσως δεν τα καταφέρουμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά σίγουρα αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να ισχύσει για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση, αλλά και να την εφαρμόσουμε. Μιλήσατε για τους μικρούς Γιώργους, τους μικροκαλλιεργητές. Σήμερα δυστυχώς υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία στην κοινωνική πολιτική. Και η διοίκηση και στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία. Οι διοικητικές αρχές ε, ε, επιβάλλουν πολλές ε, γραφειοκρατικές και ελεκτικές απαιτήσεις. Έχουν μικρές εκτάσεις αυτοί οι μικροκαλλιεργητές και το καθεστώς ελέγχου είναι πολύ δαπανηρό. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο καλύτερης υποστήριξης ε, ε, αυτών των γεωργών. Να εφαρμόσουμε μεν τον έλεγχο, να μην εκφεύγουν το έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε σε αυτές τις μικρές καλλιέργειες, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, κάποιες δυνατότητες για ανάπτυξη. Είτε ε, για έξω γεωργικές δραστηριότητες, στον ίδιο τόπο, χωρίς να χρειάζεται να μετακομίσει ο Γιώργος χωρίς να χρειάζεται να αφήσει το χωριό του για να πάει σε μεγαλύτερη πόλη είτε αν κάποιοι τέτοιοι μικροκαλλιεργητές αποφασίσουν για έξω γεωργική δραστηριότητα να δώσουμε δυνατότητα στους ενδιαφέροντα να κάνουν γεωργική δραστηριότητα να τη συνεχίσουν. Περισσότερα κονδύλια για τη δραστηριότητα για τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ανταγωνιστικής γεωργίας. Αναφερθήκατε και στην ευημερία των ζώων. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από τότε που σχεδόν ο άνθρωπος αποφάσισε να εκτρέψει ζώα για την κατανάλωση, για την ανθρώπινη κατανάλωση, ουσιαστικά αυτά τα ζώα βρίσκονται σε εχμαλωσία και μάλιστα σε εχμαλωσία υπό αφύσικους και απάνθρωπους. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε προβληματισμούς για, για τα πουλερικά στις στοιχείες κλωβών. Θέλουμε τουλάχιστον τα κλοβιά αυτά να είναι για τις οτόκες όρνηθε κάπως πιο άνετα. Σίγουρα θα πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις διατάξεις για την ευημερία, αλλά να εξασφαλίσουμε και αρκετό χρόνο για να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές. Και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Αναφερθήκατε στα θέματα των κλωβών, στις στοιχείες κλωβών. Εκεί πραγματικά έχουμε πρόβλημα ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά εξαιτία των διαφορετικών διατάξεων για, αυτά, για αυτές τις στοιχείες. Το θέμα όμως ε, είναι το σύστημα άμεσων ενισχύσεων δεν δημιουργεί στρέβλωση ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και αυτό. Και από τη στιγμή που δίνουμε μάχη για τις συστοιχής κλοβών, με την ίδια αποφασιστικότητα θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αρθούν και άλλα στοιχεία της τρέβλωσης του ανταγωνισμού και να το κάνουμε από κοινού και να δεσμευτούμε ότι θα συνεργαστούμε στενά για να αρθούν πραγματικά όλοι οι φραγμοί στον α, θεμητό ανταγωνισμό. Αναφερθήκατε και στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. αν στην Ευρώπη έχουμε κάποιου φόβου και ανησυχίε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τι απειλέ κατά το περιβάλλον, τι ε, απειλέ κατά τη βιοπικιλότητα για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού και θέλουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη διακριτική ευχαίρεια και ελευθερία επιλογή για τα θέματα αυτά, είμαστε συνεπεί Α κάνουμε το ίδιο και για τις εισαγόμενε ζωοτροφές που είναι γενετικώς μεταλλαγμένες. Και να κάνουμε το ίδιο και με τις εισαγωγέ τροφίμων από άλλε περιοχέ του κόσμου που παράγονται είτε με γενετικά τροπημένες καλλιέργειες είτε πρόκειται για κρέας ζών που ε, τρέφεται με μεταλλαγμένες ζωοτροφές. Αν είμαστε συνεπείς, συμφωνώ. Συνεπείς σε όλα. Γιατί αν τώρα ασχολούμαστε περισσότερο με το θέμα του φόβου για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που καλλιεργούνται στην Ευρώπη και ξεχνάμε τε, τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές ή τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που εισάγουμε, διαρωτώμε, εξυπηρετούμε έτσι το συμφέρον των καταναλωτών μας, εξυπηρετούμε το συμφέρον των γεωργών μας. Υπάρχει. Ποιο, ποιο συμφέρον εξυπηρετούμε στην περίπτωση αυτή. Έχω λίγο χρόνο ακόμη κύριε Πρόεδρε. το θέμα του πακέτου της ποιότητας. Νομίζω θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι καταναλωτές περιμένουν ενημέρωση πληροφορίες και η παραγωγή είμαστε υποχρεωμένοι τα προϊόντα μας να είναι υψηλής ποιότητας και η παραγωγή μας να είναι ασφαλής. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις στον τομέα αυτό. Όλα αυτά δεν θα γίνουν δωρεάν. Είναι δαπανηρές διαδικασίες. Και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για το αν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2017 για το πακέτο αυτό. Αλλά νομίζω ότι η κοινή γνώμη και οι καταναλωτές δεν θα μας δώσουν τόσο χρόνο. Οπότε το σχέδιο αυτό που έχει εγκριθεί και ελπίζω να βρούμε συμβαστικέ λύσει στη διάρκεια τη Πολωνική Προεδρία για το πακέτο ποιότητα. Εγώ θα ήθελα να, να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Πάντω, το κόστο του πακέτου ποιότητα ε, θα επιρρηθεί σε δύο πλευρέ. Στου γεωργού και στου καταναλωτέ. Α μην έχουμε ψευδεστήσει ότι αυτέ οι δύο πλευρέ θα υπομισθούν το βάρο αυτού του πακέτου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θέση του γεωργού και του μεταποιητή στην αλυσίδα τη τροφική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό χρόνια ολόκληρα. Είχαμε και ομάδα υψηλού επίπεδου για την ατροφική αλυσίδα. Τώρα υπάρχει επιτροπή υψηλού επίπεδου. Και θα ήθελα να σα πω το εξή. Και από την πρώτη και τη δεύτερη έκθεση, εγώ δεν έμεινα πλήρω ικανοποιημένο. Γιατί εμείς ε, περιμένουμε λύσει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη θέση του Γεωργού, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη θέση του μεταπίτη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί φοβούνται να επηρεάσουν το επίπεδο εμπορίου. Και σε ό,τι αφορά το επίπεδο του εμπορίου και τις ε, επιρροής που έχουν οι μεταποιητές, ε, οι μεταποιητές επί των γεωργών, ε, είναι δύσκολη η πολιτική να ταράξουν αυτή την ισορροπία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε όλοι από κοινού θάρρος και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπεροχή του εμπορίου επί των ε, μεταποιητών και επί των ε, γεωργών. Η διανομή είναι ισχυρότερη, το εμπόριο είναι πολύ ισχυρότερο και από τους γεωργούς και από τους μεταποιητές. Επίσης, ε, για το πακέτο του γάλακτος και τη μεταρρυθμίση της γαλακτοκομικής αγοράς. Μετά από επισκόπηση της κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και μετά την κρίση του γαλακτοκομικού τομέα του 2008-2009, αποφασίσαμε να κάνουμε μία ανάλυση τη αγορά του γαλακτοκομικού τομέα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για το 2010-2012. Από ό,τι ξέρω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε προτάσεις ε, για την ανάγκη αξιολόγησης της αγοράς γαλακτοκομικού τομέα μέχρι το 2012. Ε, σε ό,τι φορά την αντικατάσταση των ποσοστώσεων από συμβάσεις, για τους οποίους μάλιστα δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν νομίζω ότι αυτή η αντικατάσταση είναι αρκετή. Και ως εκπρόσωπος χώρας με μεγάλες ποσοστώσεις και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της γαλακτοκομικής παραγωγής, θα έπρεπε να είμαι ο πρώτος υπέρμαχος της κατάργησης των ποσοστώσεων και της ελεύθερης εμπορίου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι χωρίς ποσοστώσεις οι Πολωνοί κτηνοτρόφοι θα αυξήσουν την παραγωγή τους. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολύ εύκολα μπορούν να ξαναπέσουν την παγίδα της υπερπαραγωγής αν τους αφήσουμε ελεύθερους. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου έχουμε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την κρίση του 2009. Ας παρατηρήσουμε πρώτα την αγορά. Και αν πραγματικά το 2012 διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαταράξεις, τότε να εφαρμόσουμε το σχέδιο. Αν υπάρξουν όμως διαταράξεις, θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε από την νομοθετική πρόταση. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στην τροφική αλυσίδα και την υπεροχή του εμπορίου του, σε αυτή την αλυσίδα. Τώρα, αν αντί για ποσοστώσεις έχουμε συμβάσεις μεταξύ κατακόρυφες συμβάσεις παραγωγής, τότε διαρωτώ με αν στην Ευρώπη διαμορφωθούν τρία-τέσσερα ολιγοπόλια ε, με την ε, επιρροή συγκεκριμένων ομίλων και οπότε στα πλαίσια συγκεκριμένου τέτοιου, συγκεκριμένου τέτοιου λιγοπολίου, ποια πιστεύατε θα είναι η κατάσταση του Γεωργού ή του κτηνοτρόφου. Θα είναι καλύτερη ή χειρότερη. Γιατί σήμερα στην πρόταση έχουμε 3,5% περιορισμό στην ε, πανευρωπαϊκή αγορά. Και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση, αλλά δεν ξέρω θα ειναι καλυτερη η χειροτερη γιατι σημερα στην προταση εχουμε 35 περιορισμο στην πανευρωπαικη αγορα και ειναι ενδιαφερουσα αυτη η προταση αλλα δεν ξερω θα αν θα είμαστε σε θέση να την ε, κρατήσουμε και να την εφαρμόσουμε. Δεν μπορώ να το προβλέψω ακόμη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός και θα ήθελα να πείτε στους Γερμανούς Γιώργους ότι δεν είμαι, υπέρ, δεν είμαι, δεν είμαι κατά της απελευθέρωσης της αγοράς του γαλακτοκομικού τομέα, αλλά είμαι ρεαλιστής και βλέπω ότι υπάρχουν πολλές απειλές για την αγορά αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά όλες τις περιστάσεις πριν λάβουμε μια απόφαση. Ο κύριος Ολενίτσακ αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για τις εμπορικές σχέσεις. Αυτό αφορά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Μερκοσούρ, τις συμφωνίες Μερκοσούρ, αλλά αφορά και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Εμείς ε, γνωρίζουμε τη Ρωσία, είμαστε γείτονες, αλλά όχι μόνο λόγω γειτονίας. Γνωρίζουμε τη Ρωσία και πιστεύω ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, δυνάμεθα και επιθυμούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη. Η Ρωσία είναι εταίρος με τον οποίο δεν συζητούμε μόνο με την ε, εκφώνηση διακηρύξεων δηλώσεων ή με την ανταλλαγή αλληλογραφίας. Η Ρωσία και οι πολιτικοί της ε, προτιμούν άμεσες διαπραγματεύσεις και όχι μέσω επιστολών. Και νομίζω ότι οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα αυτή την ε, διάθεση των Ρώσων στα πλαίσια της κρίσης με το κολοβοκτηρίδιο. Γιατί αυτοί πρωτοστάτησαν στις ε, διαπραγματεύσεις και στη συμφωνία με την Ρωσία. Και η αρμόδιοι επίτροποι ουσιαστικά υπέγραψαν αυτή τη Γενική Συμφωνία. Αλλά χρειάζονται και επαφέ, χρειάζονται συνομιλίε και των επιτρόπων αλλά και των συγκεκριμένων μεμονωμένων χωρών. Πάντω, διαπιστώνουμε πραγματικά πόσο διαφορετικά είναι τα ελεγκτικά συστήματα που έχουμε στι διάφορε χώρε. Πόσο διαφορετικά λειτουργούν αυτά τα συστήματα ελέγχου στις χώρες. Και δεν με εκπλήσει που κάθε εισαγωγέας προϊόντων ευρωπαϊκών θέλει να ξέρει από ποια περιοχή και από ποιο ελεκτικό σύστημα πέρασε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, και, και έχει το δικαίωμα ο εισαγωγέας να θέτει αυτές τις ερωτήσεις και να λαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος. Αν τώρα τη συμφωνία και τα έγγραφα που έχουμε υπογράψει με την Ρωσία είναι ίδια για όλους, τότε ή και η θέση της Ρωσίας απέναντι σε διάφορες χώρες δεν θα έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό, εκτός από τα έγγραφα, θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στις συζητήσεις, στις επαφές με τους Ρώσους ε, πολιτικούς. Αν θεωρούμε φυσικά ενδιαφέρουσα για την Ευρώπη την ρωσική αγορά. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η ρωσική αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως κυρίες και κύριοι να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, ήταν πολύ θετική η εντύπωσή μου από τη σημερινή συζήτηση. Α, ο κύριος Μπαμπουχόφσκι μου επισήμανε το πρόβλημα του κάπινγκ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να στραφούμε κυρίως σε τρία στοιχεία της μεταρρύθμισης κοινή γεωρικής πολιτικής και να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Συμφωνήσαμε ότι οι επόμενες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να απλουστεύσουν την κοινή γεωρική πολιτική. Αναφέρθηκα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά δυστυχώ το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν προβλέπει με πολλές απλουστεύσεις. Και όταν βλέπουμε τις προτάσεις του Νοεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά, πολλές προτάσεις για απλούστευση της Γεωργίας. Υπάρχει και το θέμα του πρασινίσματος. Αλλά και το θέμα του πρασινίσματος ουσιαστικά μιλάει για εφαρμογή των προδιαγραφών που υιοθετήσαμε. Και είπαμε πολλαπλή συμμόρφωση, cross compliance για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση. Εφαρμόζουμε όλη αυτή την ε, πολλαπλή συμμόρφωση. Έχουμε εντάξει στο εσωτερικό δίκαιο όλη την οδηγία για το περιβάλλον. Θα πρέπει να ελέγξουμε αν ε, στα πλαίσια των ε, θετικών γεωργικών πρακτικών εφαρμόζονται από όλες χώρες αυτές. Είχαμε, έχουμε ήδη τρία μόνο στοιχεία που αν πραγματικά τα εφαρμόσουμε πλήρως η κοινή γεωργική πολιτική ήδη θα ήταν πιο πράσινη. Ακόμη και αν εξετάσουμε αυτή την εφαρμογή των τριών στοιχείων. Και τα επόμενα ε, στοιχεία του πρασινίσματο θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα και να έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα του κάπινγκ και τη σταδιακή μείωση. Το θέμα του ανώτατου ορίου δηλαδή και τη σταδιακή μείωση. Και αν ε, είχαμε λιγότερα κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις και της, ε, των ενισχύσεων για την παραγωγική τιμότητα και αν δίναμε περισσότερα κονδύλια για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τότε το πρόβλημα του κάπινγκ, του ανατορίου δεν θα ήταν τόσο φλέγον όπως σήμερα. Ούτε θα ήταν τόσο εξόφθαλμο και κραυγαλαίο. Το τρίτο στοιχείο η πρόταση για τον ενεργό γεωργό στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ο ενεργός γεωργός, ο δραστήριος γεωργός είναι ο γεωργός που σκέφτεται και την ανάπτυξη της γεωργικής του εκμετάλλευσης, που σκέφτεται και την ε, διαμόρφωση ε, της ανταγωνιστικότητάς του απέναντι σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ε, ένας ε, παραγωγός που σέβεται τις ε, συνθήκες και τις διατάξεις εσωτερικής αγοράς είναι δίκαιος και θα πρέπει να τη χάνει και κάποιες οικονομικές επιβράβευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για το πάθος με το οποίο απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και που μας αποσαφηνήσατε τον προσανατολισμό της Πολωνικής Προεδρίας, της δεσμεύσεις, η ατζέτα και κυρίως ε, τα ευαίσθητα θέματα. Τώρα θα κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Υπουργό και κατόπιν θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Grazie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 No, Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι θα αφήσουμε κατά μέρος το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Θα το αναβάλουμε. Θα αναβάλουμε την ψηφοφορία για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών για την ευθυγράμμιση με τη συνδίκη τη Λισαβόνας. Το αναβάλουμε γιατί πρέπει να έχουμε ένα περαιτέρω προβληματισμό μεταξύ μας ε, και για να βελτιώσουμε τη στρατηγική της ε, Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου έναντι της Κομισιόν και του Συμβουλίου σε σχέση με το θέμα της εφαρμογής της ευθυγράμμισης μάλλον στη συνθήκη της αγώνας Το αναβάλουμε. Λοιπόν, το σημείο 9. Α περάσουμε στην πράσινη βιβλίο, σημείο 10, από τι προσκλήσει ευκαιρίε προ ένα κοινό πλαίσιο στρατηγική για τη χρηματοδότηση τη έρευνα και τη καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, συντάκτη ε, είναι ο κύριος Τζοβάνι Λαβία. Του δίνω το λόγο αν επιθυμεί να πει κάτι πριν από τη ψηφοφορία. Όχι, δεν θέλει να πει τίποτα. Επομένω, α περάσουμε στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλη την ε, κάρτα Τη ψηφοφορία. και αν ναι, σας καλώ να ψηφίσετε δια τη ηλεκτρονικής οδού. Ιστολία τιμή. Ξεκινάμε λοιπόν με το συμβιβαστική πρόταση 1. Άρχεται η ψηφοφορία για το συμβιβασμό υπαρθμών 1. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην τροπολογία υπαριθμών 4. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. λήξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 4. Απορρίπτεται. Προσοχή, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία ψήφος παραπάνω για το ΕΛΚ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ας περάσουμε στην τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία για την υπαριθμόν 6. Τροπολογία, λήξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 6. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία υπερθμόν 6. Πρέπει να ψηφίσουμε και για την υπερθμόν 5. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε την ψηφοφορία για την υπερθμόν 5 Ντάντσιλα. Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Λήξη ψηφορία. Εγκρίνεται. Και αυτή η τροπολογία. Ας περάσουμε στην υπαριθμό 7. Νικολέσκου. Άρχεται η ψηφορία για την 7. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την υπαριθμό 8. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Για την 8 και απορρίπτεται. Τροπολογία είναι απάξας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 9. Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάλι έχουμε μία ψήφο συν του ΕΛΚ. Προσοχή. Μία παραπάνω ψήφο. Συνεχίζουμε. 10. Ψηφίζουμε την υπερθυμόν 10. Έχουμε ακόμα μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ. Προσοχή. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας για το 10 εγκρίνεται. Attenzione Λοιπόν, ε, ελέγχουμε. Συνεχίζουμε. Ας περάσουμε στην υπαριθμόν 11. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 11. Votazione chiusa. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία για το 13. Απορρίπτεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό υπερθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία για το συμβιβασμό 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφορία 18. Νικολέσκου. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Άρχεται η ψηφοφορία για την 19η τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, άρχεται η ψηφορία για το συμβασμό 3. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 23η. Τροπολογία. Άρχεται η ψηφορία. Για την 23η τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 Νικουλέσκου, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Πόλσον και λοιπή. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Άρχεται ψηφοφορία. Το έχουμε την ίδια πλειοψηφία, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Ντόρφμαν. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 29, Νικουλέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Και 30. Ψηφίζουμε την 30 τροπολογία. Απορρίπτεται. Και ας ψηφίσουμε τώρα επί της ε, έκθεσης, επί της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφορία, πέρας, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Στον εισηγητή, μπράβο. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 11 τη σημερινής διάταξης. Και πάλι εδώ έχουμε ψηφοφορία. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Μαρόκου αμοιβαία απελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και τα λεφτικά προϊόντα. Εδώ έχουμε η υιοθέτηση της γνωμοδότηση του κυρίου Φοντάνα. Όπως γνωρίζετε, την έκθεση αυτή πρέπει να εκφράσουμε μια γνωμοδότηση για την, για την Επιτροπή. Τα παρουσιάστηκαν δύο τροπολογίες από μέλη που δεν συμφωνούν με αυτή την πρόταση θα ψηφίσουμε πρώτα αυτές τις τροπολογίες. Αν απορριφθούν, τότε θα ψηφίσουμε το σύνολο τη γνωμοδότηση του εισηγητή. Αν και αυτή απορριφθεί, η Επιτροπή Άγκρη δεν θα στείλει καμία γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ίντα. Έτοιμοι. Λορέντσο, αν δεν θες το λόγο, να προχωρήσουμε γρήγορα στην ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε την πρώτη τροπολογία. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ας περάσουμε στην ψηφορία της έκθεσης του εισηγητή. Ψηφίζουμε την έκθεση Φοντάνα. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου, λοιπόν, μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας στην Επιτροπή Ίνταλ. Και ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, σημείο 12. Τη ημερησία διάταξη πώ θα προσπαθήσει σπατάλη τροφίμων, στρατηγικέ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τροφική ελσίδας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είναι ο κύριο Λιβατόρα Καρόνα. Η αποτελεσματικότητα τη τροφική αλυσίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα. Όπω ξέρετε, το 1 τρίτο των τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή δαπανάται κυρίω σε βιομηχανοποιημένε χώρε και αυτό αποτελεί μια τεράστια σπατάλη πόρων και παράγει τεράστιε ποσότητε εκπομπών. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτή την πρόταση γνωμοδότηση. Να σα ενημερώσω επίση ότι Έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την οποία η έκθεση αυτή θα είναι αποκλειστικά της, για αυτό το λόγο θα είναι αποκλειστικά δική μας η έκθεση αυτή, δεν θα υπάρχουν ε, το άρθρο 50 που έρχεται εδώ. Έτσι λοιπόν ο κύριος Καρόλ έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα, γιατί ήδη έχει διανεμηθεί το άγγραφο συναδέλφους. Η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας ε, γεννιέται από μία απέτηση να ε, επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα της πατάλης των τροφίμων, ένα θέμα που δυστυχώς εδώ και καιρό έχει υποτιμηθεί και που κατά τη ε, διάρκεια του χρόνου, με το πέρασμα του χρόνου, πήρε μια πολύ σημαντική διάσταση. Τα επίπεδα της πατάλης ε, τροφίμων, έτσι όπως εκτιμούνται, είναι τόσο μεγάλο που λέμε ότι δεν βρισκόμαστε μόνο ενώπιον σε ένα πρόβλημα ηθικού ε, χαρακτήρα, αλλά είναι και ένα πραγματικά οικονομικό ζήτημα με πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες και για το περιβάλλον τα στοιχεία πραγματικά είναι ανησυχητικά. Σύμφωνα με μια μελέτη της ΦΑΟ, το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται κάθε χρόνο στον κόσμο και για την κατανάλωση του ανθρώπου χάνεται ε, και σπαταλάτε μιλάμε περίπου για 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων που πάνε στα σκουπίδια. Στην Ευρώπη όπως ε, και στην Βόρεια Αμερική έχουμε σπατάλη 115 κιλά τροφίμων ετσίως ανάτομα ενώ ε, στην Αφρική 11 κιλά μπορούμε να πούμε ότι τα τρόφιμα ε, που κάθε χρόνο σπαταλούνται ισοδυναμούν με το ίμιση της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών. Η Ευρώπη είναι, ένα από, είναι μία από τις περιοχές του κόσμου όπου γίνεται περίπου το 50% αυτής της σπατάλης. Είναι πλέον οξύ αυτό το φαινόμενο. Αν ε, σε όλο τον κόσμο υπήρχαν ε, αυτοί οι ρυθμοί, θα χρειαζόμασταν τρει πλανήτε για να παράγουμε την απαραίτητη ποσότητα τροφίμων. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον ενό παγκόσμιου φαινομένου το οποίο αφορά όλα, ε, όλες τις τους κρίκους ε, τη τροφική ολυσίδα, ξεκινά από τον αγρό και φτάνει μέχρι τον καταναλωτή. Το φαινόμενο αυτό αφορά κυρίως τις ε, πιο αναπτυγμένες χώρες, αλλά ω ένα βαθμό και τι αναπτυσσόμενες. Αν ε, για τις πρώτες το πιο σχετικό τμήμα της πατάλης βρίσκεται στα τελευταία στάδια της αλυσίδας, δηλαδή από τη διανομή στην κατανάλωση, για τι αναπτυσσόμενες χώρε. αυτή η πατάλη τη βλέπουμε κυρίως στο στάδιο τη παραγωγή τη εσοδιάς ε, και της διανομής επειδή δεν υπάρχουν πρεγμένες ε, τεχνολογίες ε, και δυνατότητες αποθήκευσης ή υποδομές μεταφοράς. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι όλα αυτά έχουν ένα κόστος Πέρα από το οικονομικό κόστος υπάρχει και ένα σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος περίπου 90 εκατομμύρια ε, τόνοι τροφίμων ε, που καταλήγουν στα απόβλητα κάθε χρόνο παράγουν 170 τόνους διεξουδίου του άνθρακα. Ε, πέρα και από άλλες σκέψεις που ουσιάζονται στην έκθεση πρωτοβουλίας ε, και αυτά μας κάνουν να πούμε ότι θα πρέπει η σπατάλη τροφίμων ε, να καταστεί προτεραιότητα στο ιστορικό της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντα και γι' αυτό είναι σημαντικό η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια στρατηγική και συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσουν την τάση αυτή θέτοντας ε, ένα πολύ φιλόδοξο στόχο που είναι όμως εφικτός μέχρι το 2025 να μειωθεί σημαντικά το φαινόμενο αυτό να καταστούν υπεύθυνοι όλοι οι πρωταγωνιστές της αλυσίδα, ε, ξεκινώντας από τον αγρό μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή. Γι' αυτό προτείνουμε και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης όπου θα συμμετέχουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, αλλά ακόμη και μεγάλες ε, αγροτικές οργανώσεις και η βιομηχανία, να υπάρχει ενημέρωση για τις συνέπειες αυτής της φαντάλης τροφίμων. Να προωθήσουμε λοιπόν ε, έναν ε, πολιτισμό που προσανατολίζεται, μια κουλτούρα που προσανατολίζεται προ ένα πιο βιώσιμο τρόπο κατανάλωση. Σε διάφορα κράτη τη Ένωση υπάρχουν εμπειρίε που προωθούνται από ενώσει και από θελοντικέ ομάδε που υλοποίησαν ε, προγράμματα κατά της πατάλης των τροφίμων. Όλα αυτά οδήγησαν ε, σε ένα σύστημα αφαφλού Αντί, όμως, αντί να μειώνεται δηλαδή η σπατάλη των τροφίμων, μάλλον σε ένα ενάρετο σύστημα, με συγχωρείτε, οδήγησε, ε, αντί να κατασφαλίζονται τα τρόφιμα, δίνονται σε απόρου και σε ανθρώπου με οικονομικέ δυσκολίε. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή μια νομοθετική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το ζήτημα αυτό και ε, ξεκινώντας ε, και από το ότι δεν ε, υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τις σπατάλη των τροφίμων. Έτσι λοιπόν θα επιθυμούσαμε η Κομισιό να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση που να προσδιορίζει την τυπολογία της σπατάλης των τροφίμων. Και ετέλει, αλλά εξίσου σημαντικό, επισημαίνουμε στην έκθεση να διακηρυχθεί το 2013 ως το Ευρωπαϊκό Έτος κατά τη σπατάλης των τροφίμων. προκειμένου να υπάρξει ανανεωμένη δέσμευση ε, όλων των ευρωπαϊκών θεσμών για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας ε, για οποιοδήποτε ερώτηση. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Καρόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Καλό λοιπόν ε, όλους τους κοιόδης να εργαστούν εντατικά για το θέμα αυτό, το οποίο θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Τώρα, ξεκινάμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η σπατάλη των τροφίμων είναι σοβαρότερο πρόβλημα από ό,τι μέχρι τώρα νομίζαμε. Γύρω στο 1 τρίτο των τροφίμων που κουβαλάνε στο σπίτι οι καταναλωτές στη ΣΥΠΑ πετάγεται. Και όσο πιο αργά συμβαίνει αυτό στην αλυσίδα, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, λέει και ο εισηγητής, ε, βρίσκεται στη μεταφορά και την αποθήκευση και είναι όντως ε, σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να συνεισφέρουμε στο να έχουμε ένα σταθερό ε, σύστημα το οποίο θα λειτουργεί. Αλλά στις στοχές χώρες ούτως ή άλλως πετάνε πάρα πολύ λίγα ε, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση νομίζω. Όσον αφορά δε τη σπατάλη της ενέργειας, το αντιμετωπίσαμε αυτό, το είχαμε δει πριν από 10 χρόνια, γιατί ξέρετε τότε ήταν πολύ φτηνή ενέργεια και δεν υπήρχε κόστος και δεν μας απασχολούσε το πρόβλημα. Μετά έγινε πιο ακριβή και σήμερα βλέπουμε πως υπάρχουν προβλήματα στον τομέα αυτών. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε κάτι ανάλογο για τα τρόφιμα. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η σπατάλη. Τα τρόφιμα δεν θα είναι πλέον τόσο φτηνά όσο ήταν. Εγώ θα επιθυμούσα να έχουμε ένα πρόγραμμα ή, μπας περιπτώσει, να ξεκινήσει μια διαδικασία σκέψης όπως έγινε με την ενέργεια. Σήμερα μιλάμε για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και να λέμε με ναι, τα τρόφιμα γιατί Ξέρετε πως ε, πολλά απαιτιούνται. Ε, βεβαίως αυτό είναι δύσκολο, θα απαιτήσει χρόνο, αλλά πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Εγώ είμαι παιδί του πολέμου, με στείλανε στην Ήπεθρο ε, στους βομβαρδισμούς τότε. Ε, εκεί πέρα ζούσαμε γεωργούς που έκαναν τα πάντα και σταύρωναν το ψωμί πριν το φάνε. Για μένα αυτό είναι ένα σύμβολο. Για το ότι πρέπει να σεβόμαστε το ψωμί που τρώμε. Πρέπει να προσέξουμε να δούμε λίγο. Να ξαναδούμε τι γινόταν ε, εκείνες τις εποχές. Γιατί αν σκεφτούμε τι κοστίζει ένα κιλό στάρι ή κρέας ή οτιδήποτε για να παραχθεί. Ε, εντάξει, είναι κάπως ε, περιορισμένο το οικονομικό κόστος, αλλά είναι μεγάλο το περιβαλλοντικό κόστος. Και αυτό ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε. Και όχι τόσο την οικονομική σκοπιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πόλσον. Άλβορτ, παρακαλώ. Και μετά ο κύριος Λαβιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Στηρίζω την πρόταση το 2013 να είναι το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της πατάλης τροφίμων. Το να ενημερώσουμε για αυτό το θέμα είναι σημαντικό και αποτελεί ένα κλειδί. Καθώς η τροφική αλυσίδα είναι παγκόσμιο ε, φαινόμενο πλέον. Το θέμα δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά να συνδεθεί με την ασφάλεια των τροφίμων και την αναπτυξιακή πολιτική και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο κόσμος περισσότερο στα αποφάγια τα πετάει ε, στο σκουπιδέντε και αλλά βεβαίως χάνονται απαράδεκτες ποσότητες σε κάθε φάση της τροφικής αλυσίδας και οι καταναλωτές είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Εγώ θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το ποια μέτρα πέρα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση μπορούν να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο σε όλες τις ε, φάσεις αλυσίδας. Χρειάζονται βεβαίως μαθήματα ε, εκπαίδευσης ε, στα τρόφιμα και πρέπει βεβαίως να δούμε και τις πατάλοι πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα κατόπιν. Ο ορισμός θα πρέπει να εναρμονιστεί έτσι ώστε οι σχετικές εκστρατείες ε, και καμπάνιες να είναι συνεκτικές και αποτελεσματικές. Και ορίζω βέβαια συμπερίληψη αυτής της σύστασης. Τρίτον, ο στόχος του να μειωθεί η σπατάλη στο μισό μέχρι το 2025 δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενημέρωσης. Πρέπει να δούμε πρακτικά μέτρα συσκευασίας και σήμανσης και Τώρα να ξαναμοιράζονται τα απόλυτα ε, τρόφιμα τα οποία είναι ακόμα βρόσιμα σε ανθρώπους με περιορισμένα μέσα. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου μπορεί ακόμα η Γεωργία να παίξει ένα ανθρωπιστικό ρόλο. Αντιμετωπίζοντα ταυτόχρονα ζητήματα ασφάλεια τροφίμων και κακή διατροφή στην Ευρώπη. Καλωσορίζω τη γενική θέση του εισηγητή και η έκθεση αυτή θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα πω η καταπολέμηση τη πατάλη αυτή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ευχαριστώ. Ονορεύολε Λαβία. Λαβία και κατόπιν Μάρτιν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Καρόνα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε μας αυτό το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Πιστεύω ότι ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση και που αναφέρει ο κ. Καρόνα θα πρέπει να μας προβληματίσουν το ότι 179 κιλά ε, τροφίμων καταστρέφονται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής ε, είναι ε, ένα στοιχείο που δεν αφορά μόνο τον τελικό καταναλωτή αλλά όλον το γεωπιστικό τομέα από τον αγρό μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ακόμη περισσότερο όταν πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις ε, της ε, αύξησης του πληθυσμού στη γη μας δείχνουν ότι θα έχουμε επιπλέον ε, δύο δισεκατομμύρια καταναλωτές και δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε αν δεν αυξήσουμε την παραγωγή και υπάρχει και ανταγωνισμός ε, σε σχέση με άλλους παραγωγικούς τομείς, το χάρη, σκέφτομαι το νερό που είναι απαραίτητο για την αγροτική παραγωγή. Ε, έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την έννοια της χρήσης και της μέγιστης μείωσης της πατάλης των τροφίμων και της βέλτιστης χρήσης των γεωπιστικών προϊόντων ε, στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών στρατηγικών που πρέπει να εγγυηθούν ε, τη διατροφική ασφάλεια, την επιστημιστική ασφάλεια ε, παγκοσμίω στο μέλλον. Έτσι λοιπόν ε, να πρέπει να ζητήσουμε έντονα από την Κομισιόν να διατυπώσει κάποιες προτάσεις γιατί όσο περισσότερο το σκεφτόμαστε το θέμα αυτό τόσο πιο πολλές ιδέες μας έρχονται στο νου για μικρές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να μειώσουν αυτή τη μεγάλη ποσότητα ε, των τροφίμων που οδηγούνται στα σκουπίδια ή που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν ε, οι κανόνες για την θεσία, η πρόταση για μερομηνία λήξης του προϊόντος ε, για την πώληση και για την τελική χρήση, όπως και τόσες άλλες προτάσεις ε, θα μπορούσαν ε, να διατυπωθούν και θα μπορούσαν να γραφούν στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο να μειώσουμε τη σπατάλη και να δοθεί μια νέα προσοχή στα τρόφιμα πιθανότητα σε μία περίοδο φθονίας ε, το χάσαμε αυτό, αλλά έτσι όπως μας υπενθύμισε και η συνάδελφος Πόλσεν, σε μία περίοδο έλλειψης αποκτούν μεγαλύτερη αξία, και όπως έχουν σήμερα πολύ μεγάλη αξία για όλες τις χώρες, ε, όπου οι πληθυσμοί τους δεν έχουν επαρκή τρόφιμα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα, ευχαριστώ Μάρτιν Όσλιν και, κατόπιν und σας ευχαριστώ για την έκθεση και τις προτάσεις που έγιναν. Όλες καλές. Να υπενθυμίσω βεβαίως πως πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε με κανονισμό είναι αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Πρέπει να πω πως πολλοί δεν ξέρουν την έκταση της πατάλης. Γιατί αυτό σχετίζεται με το ότι τα τρόφιμα δεν έχουν πλέον καμία αξία. Δηλαδή, δίνουμε τόσα λίγα λεφτά, ώστε καταλήγουν στα σκουπίδια γρηγορότερα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Αλλά όλοι γνωρίζουμε πως ε, πρέπει προσεχώς να ταΐσουμε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη παραγωγή. Αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να παραχθεί περισσότερο, περισσότερα τρόφιμα στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να χειριστούμε καλύτερα τις, ε, τους πόρους που έχουμε, όπως με την ενέργεια. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν νομίζω πως ε, πρέπει να κατηγορούμε τον καταναλωτή ότι τα πετάει στη σκουπίδια. Ήδη στην αλυσίδα χάνονται πάρα πολλά. Γιατί, κοιτάξτε και στα χωράφια, αν δούμε τις προδιαγραφές που υπάρχουν, αν είναι μικρές ε, και κοτόχοντρες οι πατάτες ε, μένουν στο χωράφι γιατί δεν ε, τις θέλει το σούπερ μάρκετ. Ήδη εκεί είναι το πρώτο βήμα. Και αυτά που δεν χρησιμοποιούνται στο σούπερ μάρκετ γιατί θέλουν να έχουν όλα την ίδια εμφάνιση και ποιότητα. Και αυτό πρέπει να δούμε. Εκεί είναι οι μεγάλες απώλειες. Και σε αναψώμενε χώρες είναι άλλο το πρόβλημα. Ε, εκεί πέρα χάνονται πάρα πολλά γιατί δεν υπάρχει αλυσίδα. Αποθήκευση δηλαδή, ψήξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε να μην μιλήσουμε μόνο για αύξηση της ε, παραγωγικότητα και τη οδεία, αλλά να δούμε και εντό του συστήματο πώ θα βελτίσουμε την ε, κατάσταση. Αυτά είναι τα αποφασιστικά συστήματα και άρα νομίζω πως υπάρχει ακόμα μεγάλη δυνατότητα στο μέλλον να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τα τρόφιμα. Και να ξέρουμε το τι γίνεται βεβαίω ε, από πλευράς σπατάλης. Πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από εκκλήσεις, συγκεκριμένα μέτρα. Και ελπίζω να α, γίνει κάτι και όχι μόνο να αυξάνεται η εισοδιά, η αποδοτικότητα. Ευχαριστώ Μπρίτα Ρήμερς και μετά Μαγκίνες. Ευχαριστώ με την έκθεση αυτή να ε, αντιμετωπίζουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ευημερία, σχετίζεται με την πολιτική σταθερότητα σε κάποιες χώρες που εμποδίζουν το να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες επιμελητίας. Οπότε θα πρέπει με μέσα πολιτικά να σταθεροποιήσουμε την ε, κατάσταση για να μην υπάρχει πλέον ε, σπατάλη στο χωράφι. Αλλά είναι μια γενικότερη ε, οικονομική και κοινωνική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και να απευθύνουμε έγκληση στον καταναλωτή γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό χάνουμε πράγματι πάρα πολλά πράγματα αλλά θα πρέπει να έχουμε συνέστηση των τροφίμων και να κοιταχτούμε και στον καθρέφτη και να δούμε τι απαιτήσει έχουμε. Ε, αν θέλουμε να τρώμε μόνο ένα κομμάτι του κάθε τροφίμου ή να τρώμε και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία σήμερα πετάμε και δεν μας αρέσουν. Ή το βράδυ να τρώμε τα αποφάγια του μεσημεριανού. Ή κάτι που είχε μείνει από χτες. Ή από δύο προηγούμενες μέρες να φτιάχνουμε ένα καινούριο φαγητό. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα μπούμε στις συνταγές. Αλλά δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν την κάνουμε. Και εμείς μπορούμε να νομοθετήσουμε όσο θέμε, δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τις πόρους, το νερό, το έδαφος, ε, ε, αυτό να μην αφορά μόνο το γεωργό και όσοι το επεξεργάζονται, αλλά και το εμπόριο να εμπλακεί να υποχρεωθεί και ο καταναλωτής να του ξεκαθαρίσουμε το ότι γίνεται, πως έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι και θέμα εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνει πολλούς τομείς κοινωνικούς. Όλες οι επιτροπές πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Γιατί μπορούμε να το λύσουμε μόνο από κοινού. Δεν είναι μόνο θέμα γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνης. Και μετά ο κύριος Σεκέρσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το πρόβλημα είναι τρομερό. Μιλάμε... Ε, θα προτιμούσα να μιλάμε για τρόφιμο που πήγε άδικα περισσότερο παρά για σπατάλη τροφίμο, για σπαταλημένο τρόφιμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, να ανακυκλώσουμε τα απόβλητα τροφίμων. Αλλά όταν μιλούμε για σπαταλημένο τρόφιμα, σπαταληθέντα τρόφιμα, νομίζω ότι έχουμε 6 με 11 κιλά ε, για την ε, υποσαχάρια Αφρική ε, σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει ελάχιστους πόρους Θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε με την επιστηστική βοήθεια της χώρες αυτές για να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να βοηθήσουμε ταυτόχρονα και επανάπτυκτες χώρες στην υποσαχάρια Αφρική. Και εγώ ε, ξεκίν, με το σλόγγαν ότι δεν θα πρέπει να σπαταλάμε, αλλά μερικές φορές... Ε, πετάμε, τουλάχιστον να μην πετάμε φαγητό που μπορεί να καταναλωθεί, τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Και το γεγονός ότι θα ορίσουμε ειδικό ευρωπαϊκό έτος για το θέμα αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα για να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση. Και ένα άλλο ε, επιχείρημα που θα πρέπει να σκεφτούμε αφορά τα συστήματα ποιότητας μας, γιατί μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι απαιτήσει του καταναλωτή που είναι αρκετά τελειωμένης. Το θέμα είναι ότι αν επιτρέψουμε πιο ελαστικές προδιαγραφές θα έχουμε μεγαλύτερη προσφορά τροφίμων και με την επίπτωση που θα έχει στην τιμή των ε, παραγωγών περισσότερο. Ε, γιατί το θέμα του τι λαμβάνουν οι παραγωγοί και τι πληρώνουν οι καταναλωτέ δεν αναφέρεται. Το θέμα είναι πώ να βελτιώσουμε την κατάσταση για να περιορίσουμε τη σπατάλη, αλλά να δούμε και τι συνέπειε που ε, υπάρχουν από το θέμα αυτό για τους ε, διάφορους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, τους παραγωγούς, μεταποιητές λοιπά Θα το επισημάνουμε σε τροπολογίες. Πάντως η έκθεση είναι καταπληκτική και ο στόχος σίγουρα ε, αξιέπαινος και σημαντικός. Το θέμα είναι πώς θα τον υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεκέρσκι έχει το λόγο και μετά ο Άλμπερτ Ντες. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια συζητήσαμε το θέμα της μείωσης των πόρων για την δωρεάν διανομή τροφίμων στους απόρους. Βλέπουμε όμως ότι οι τιμές τροφίμων είναι υψηλό, υψηλές, ε, υπάρχει ανεργία, υπάρχουν εισοδήματα και έχουμε όλο και περισσότερους φτωχούς και απόρους, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μεγάλη σπατάλη. Και αυτή η σπατάλη βέβαια εντοπίζεται κυρίως σε πιο υψηλά εισοδήματα, σε πιο εύπορα τμήματα ε, του πληθυσμού, αλλά και αυτό ίσως ε, η σπατάλη οφείλεται στο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλές ε, τις τιμές και το πόσο προσιτά είναι τα τρόφιμα. Θα, θα πρέπει να εξετάσουμε όμως και από συστημική άποψη αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε ένα κατάστημα, μια εταιρεία που για παράδειγμα θα μπορούσε να διαθέτει ε, θα μπορεί να διαθέτει σε ένα φτωχοκομείο ε, ε, τρόφιμα που είναι κοντά στο, στην ημερομηνία λήψης, αλλά, για, στην ημερομηνία αλλά ακριβώς επειδή πρέπει να πληρώσει ένα κόστος, να πληρώσει και το ΦΠΑ, δεν ενδιαφέρεται να διαθέσει ε, παραγωγικά αποτελεσματικά αυτά τα τρόφιμα που έχουν ε, σχεδόν πλησιάσει την ημερομηνία λήξη. Αυτό προτιμάει να τα πετάξει ένα κατάστημα, μια εταιρεία. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και το νομικό ζήτημα και το οικονομικό. επίση έχουμε τις ε, εμπορικές διατάξεις. Πολύ συχνά ένα υγιές τρόφιμο μόνο εξαιτία τη εμφάνισή του δεν θεωρείται επιλέξιμο για εμπορία. Αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Γιατί να μην μπορούμε να το δώσουμε αυτό το τρόφιμο που είναι απόλυτα κατάλληλο για κατανάλωση σε έναν άπορο, σε ένα φτωχό. Γιατί να το πετάμε μόνο και μόνο επειδή η εμφάνισή του δεν είναι καλή. Επίσης, σε διάφορους δημοσιονομικούς μηχανισμούς θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια αποτελεσματικά μέσα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το πολύ απαραίτητο πρώτο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. και Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ακούστηκαν. Εμένα στη ζωή μου δύο πράγματα με σημάδεψαν σε σχέση με τα τρόφιμα στα μέσα της δεκαετίας του 50 με τη γιαγιά μου στο χωράφι μαζεύαμε στάρια που είχαν μείνει πάνω στα στάχια ακόμα ε, και δεν πετάγαμε όπως καταλαβαίνετε έτσι που ζούσαμε τίποτα. Αυτό το οποίο λοιπόν ξεχνάμε με τα τρόφιμα είναι τροφή για τη ζωή τα τρόφιμα, το καταλαβαίνετε. Αλλά όταν πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ βλέπει τόσο μεγάλη προσφορά και ε, δεν έχει συνέστηση του τι είναι αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που με σημάδεψε συνέβη δεκαετία του 90. Ήμουνα με μια ομάδα από την πατρίδα μου σε ένα ταξίδι στην ε, Βραζιλία μου και πήγαμε στο Ρεσίφε ε, και φάγαμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν σιδερόφρακτο. Μας σερβιραν και γύρω γύρω είχε σειρματοπλέγματα σε μια τεράστια αγροτική χώρα γιατί οι νέοι άνθρωποι 15-16 ετών ήταν με τις πλαστικές σακούλες και μας ζητούσαν αυτά τα οποία δεν τρώγαμε να τους τα πετάξουμε στην πλαστική σακούλα. Ο δε ιδιοκτήτης του εστιατορίου ήθελε να μας το απαγορεύσει, εγώ δεν το επέρεψα. Είπα το έχω πληρώσει αυτό το φάει και θα το κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και είχαμε αφήσει ούτως ή άλλως τόσο πολύ που μπόρεσαν να φάνε άλλοι 15-16 άνθρωποι από τα αποφάγια μας. Αν δείτε δηλαδή το, το, πόσο ευγνώμονες ήταν να φάνε τα αποφάγια μας, αναρωτιέμαι καμιά φορά έτσι, με ποια ευκολία πετάμε το φαΐ. Ποτέ δεν θα φτάσουμε στο μηδέν βεβαίως, Τη σπατάλη, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Στη Γερμανία το είχα υπολογίσει. Μιλάμε για δισεκατομμύρια που πετάγονται. Μιλάμε για... Φανταστείτε, 100 ευρώ ανακάτοικο μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ήδη. Εάν συγκρίνουμε δε το ότι η Γερμανία πληρώνει 7 δισεκατομμύρια καθαρές φορές στις Βρυξέλλες, είναι, το είναι περισσότερο φαΐ πετάμε, δηλαδή σε σκουπίδια, για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί αυτή η σπατάλη. Ναι, γιατί βλέπετε πως μέχρι το 2050 πρέπει να διπλασιαστεί η παραγωγή τροφίμων, αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της μείωσης της ε, σπατάλης και με την έκθεση αυτή μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Άλμπερτ. Μάλιστα, έχουμε ακόμα τρία άτομα που έχουν ε, ζητήσει το λόγο. Στις 12 πρέπει να τελειώσουμε για να κάνουμε και τις συνεδρίες των συντονιστών. Ο κ. τους καταρχήν. Ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτόν τον προβληματισμό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι ρυθμοί της πετάλησης, τα νούμερα της πετάλησης είναι εντυπωσιακά αλλά δεν ξέρω αν η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να έχει κάποια αποτελεσματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια στρατηγική για το πώ θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτά με πρακτικέ συνέπειε. Και οι πρακτικέ συνέπειε είναι ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσω εκστρατιών, πληροφόρηση και μέσω τη εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα πρότεινα εγώ εδώ και θέλω να το προτείνω στον εισηγητή είναι να παρουσιάσουμε μια τροπολογία έτσι ώστε να αναφερόμαστε σε μια ενημερωτική εκστρατεία στο θέμα αυτό, στο ευρωπαϊκό τόσο που προτείνεται κατά της φαταλής τροφίμων που να μπορούσε να επιλεκτεί και να αφορά, παραδείγματο χάρη, να συνδεθεί και με τις εκστρατείε ε, της πρόθεση των αγροτικών προϊόντων. Ε, μια τέτοια εκστρατεία πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να έχει κάποια αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι το να φτάσουμε στους πλέον νέου, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ Νίκολσον ε, και κατόπιν Μάρκ Ταραμπέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και θα μας απασχολήσει για καιρό. Και βεβαίως δεν θα φτάσουμε ποτέ στο μηδέν της πατάλης, δεν γίνεται. Αλλά μπορούμε να, κάνουμε, να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Η δικιά μου η μνήμη φτάνει και αυτή στη δεκαετία του 50. Θυμάμαι πάντα τον πατέρα μου στο ποδήλατο που πήγαινε από το αγρόκτημά μας ε, στην ε, δημοκρατία της Ιρλανδίας που είχαν περισσότερο φαΐ και επέστρεφε με ζάχαρη και βούτυρο και μαρμελάδα, πράγματα που δεν είχαμε εμείς γιατί ακόμα είχαμε δελτία. Και τότε πραγματικά εκτιμούσε κανείς το φαΐ και το, το περίμενε, περίμενε να επιστρέψει κανείς γιατί ήταν κάτι το, το ιδιαίτερο. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω το κόσμος έχει κακομάθει γιατί έχει πολλές επιλογές η δυνατότητα δηλαδή να αγοράσουμε τρόφιμα που μάλλον είναι και φτηνά, πολύ φτηνά κατά την άποψή μου. Ε, μάλλον επηρεάζει αυτή τη συμπεριφορά. Νομίζω λοιπόν πως η Κομισιόν μπορεί να κάνει πάρα πολλά και εμείς και ε, υπάρχει στα σούπερ μάρκετ και αυτή η ημερομηνία λήξης. Ε, κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι το θεωρούν ως κάτι το απόλυτο. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ Σάββατο ε, και τα πράγματα λήγουν την Κυριακή. Τα αγοράζω, το μαγειρεύω, το τρώω και είναι μια χαρά. Αλλά πολλοί κόσμος Και νομίζω πως αυτός είναι ένας καλός τρόπος να διαθέσουμε αυτό το φαγητό. Καλό είναι να ξαναδούμε έτσι τα βασικά. Αντί για μας που έχουμε φτάσει στα υψηλά κλιμάκια. Και κάποιοι μας λένε πως ε, μπορούμε να κάνουμε θαυμάσια πράγματα και θα είναι η ζωή ωραία. Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία για συζήτηση και θα έχουμε καλέ νέες ιδέες. Αναμένω αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε Τζιν. Ο Μάρκ Ταραμπέλα θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Παύλο. Όντω η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Μπράβο Σαλβατόρε Καρόνα. Νομίζω ότι σήμερα ε, δεν σεβόμαστε το, τα τρόφιμα στο παρελθόν και με το φάσμα των πολέμων που γνωρίσαμε στην Ευρώπη, σίγουρα οι προηγούμενες γενιές, αυτές που γνώρισαν το φάσμα του πολέμου και την ε, πείνα που του συνόδευσε, ε, είναι γενιές που εξαφανίζονται σιγά σιγά. Οπότε αυτός ο σεβασμός προς το τρόφιμα έχει εξαφανιστεί. Θυμάμαι τα λόγια των, ε, του μπαμπά μου, του, του παππού μου που λέει δεν σπαταλάμε τίποτα, τρώμε το ψωμί ακόμη και αν είναι ξερό, ακόμη και αν έχει περάσει χρόνο, αλλά δεν πετάμε τίποτα. Και το θέμα της διαπαιδαγώγησης, μερικές φορές ε, λέμε ότι το σχολείο θα πρέπει να αναλάβει αυτό το θέμα, αλλά όντως ε, εκεί περνάνε 6 με 18 χρόνια πολλοί οι μαθητές. Οπότε όπως λέει η παράγραφος 9, μέσω της παιδείας και χάρη σε καλύτερη διαπαιδαγώγηση που θα γίνει μέσα από το σχολείο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά έχουμε και την ευθύνη της αγοροπιστιστικής βιομηχανίας. Μπορεί να παίξει ρόλο σε ό,τι αφορά το μέγεθος συσκευασία, γιατί πολλά ε, τρόφιμα συσκευάζονται στην ίδια διαδικασία και όταν δεν ε, τα καταναλώσουμε αμέσως και αλλάξουν χρώμα ακόμη και στο ψυγείο, τα πετάμε, ενώ εξακολουθούν να είναι βρόσιμα και κατάλληλα για κατανάλωση. Και εκεί θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τη βιομηχανία. Και το τρίτο θέμα, η πολιτική των αποβλήτων. Μερικές χώρες έχουν πολύ ε, ε, περιοριστικές πολιτικές για την διαχείριση των αποβλήτων, επεξεργασία, ε, διαχωρισμό. Ε, ίσως όμως υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ε, αναγκαστικής ε, περιοριστικής πολιτικής, όπου δίνουμε περισσότερη έμφαση στο ρηπαίνο πληρώνει και όσος παράγει περισσότερα, όποιος παράγει περισσότερα απόβλητα τα πληρώνει. Μήπως αυτό έχει σχέση με την ε, συμπεριφορά του καταναλωτή. Αυτό ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ίσως έτσι ε, μειώσουμε και τη σπατάλη τροφίμων, αλλά μειώσουμε και τα απόβλητα. Ευχαριστώ Μάρκ, ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο και ευχαριστούμε φυσικά και τον εισηγητή. Θέλω να υπενθυμίσω γιατί ήταν ε, και το μιλό της έργας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή το πώς θα αποφευχθεί σπατάλη, όχι πώς θα, γίνε, θα γίνεται η διαχείριση αυτής της ε, σπατάλης ε, και των αποβλήτων. Γι' αυτό είναι αρμόδια η Επιτροπή Τώρα θα δώσω τον ε, λόγο στον εκπρόσωπο της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ αν θέλει να μας πει κάτι και κατόπιν θα ξαναδώσουμε τον λόγο. Στον εισηγητή Επιτροπή, θέλετε το λόγο. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ευχαριστώ η Κομισιόν θεωρεί αυτή την ε, πρωτοβουλία ιδιαίτερα σκόπιμη και προσδεκτή για να αναλάβουμε δράση και να θέσουμε ως προτεραιότητα την ανάληψη δράσης κατά της πατάλης των τροφίμων. Ε, αποτελεί και αυτό μία από τις θεματικές πρωτοβουλίες για την Στρατηγική Ευρώπη 2020, η ορθή διαχείριση των πόρων. Ε, η Ευρύτα προτείνεται να δώσουμε στο θέμα αυτό είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να συμμετέχουν διάφοροι πρωταγωνιστές στη διατροφική αλυσίδα αλυσίδα από τον αγρό μέχρι τον καταναλωτή και μιλάμε και για τη συμμετοχή των ΜΚΟ, ε, τη εκπαιδευτική κοινότητα. όλα αυτά αναφέρθηκαν, αλλά Επίση, αυτό είναι απαραίτητα για να ευνοήσουμε και τι συνέργειε μεταξύ διαφορών πολιτικών και δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να συνδράμουν στο στόχο τη μείωση ε, τη φατάλη των τροφίμων. Η προκαταρκτική μελέτη που ζητείται από την Επιτροπή και που αναφέρεται στην ε, έκθεση του κ. Καρόνα ε, αφορά μια πρώτη διάγνωση για τη σημασία του προβλήματος και τους παράγοντες ε, πρόκλησης. Πρόκειται για μια πρώτη αξιολόγηση ε, και η ανάληψη πρωτοβουλειών ουσιαστικά μας οδηγεί σε μια πρώτη ανάληψη δράσης από τις ευρωπαϊκούς θεσμούς για να κατανοήσουμε καλύτερα και να εποπτεύσουμε την εξέλιξη του φαινομένου, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένε ε, αμφισημίες, κυρίως ό,τι αφορά την επισήμανση που οδηγούν ε, το σχάρι ε, και στην κατηγοριοποίηση ενό τροφίμου ως απόρριμα αλλά εξακολουθεί να είναι βρόσιμο οι απώλειε στον ίδιο τον αγροτικό τομέα δεν έχουν διαρευνηθεί. Λέγεται στην έκθεση, αλλά είναι ε, αλήθεια ότι δεν έγκυται εκεί το πρόβλημα. Κυρίως ε, το πρόβλημα βρίσκεται στις βιομηχανοποιημένες χώρες ε, προς το πάνω μέρος της τροφικής αλυσίδας. Σε ό,τι αφορά παρόλα τα όρια τους, αυτές οι προκαταρτικές μελέτες μας δείχνουν το μέγεθος και τη σημασία του προβλήματος και επίσης ε, την πρόλευσή του και τις προσπάθειες ε, ε, που γίνονται δεσμεύουν ε, ένα σύνολο πρωταγωνιστών και άπτονται έναν, ε, ενός αριθμού διάφορων πολιτικών που υποστηρίζουν ή επηρεάζουν τις προσπάθειες των διάφορων συμμετεχόντων. Έτσι λοιπόν, σε ένα πρώτο χρόνο πρέπει να έχουμε ένα συντονισμό πολιτικών και να ασχοληθεί και δια Κομισιόν. Ε, ε, μου ζητήσατε να είμαι σύντομος, έτσι λοιπόν δεν θα αναφερθώ στις ε, τρέχουσες πρωτοβουλίες. οι οποίες ουσιαστικά συμφωνούν με τον προσανατολισμό που αναφέρεται εδώ. Έτσι λοιπόν, ε, εμείς συμφωνούμε με όσα λέει ο εισηγητής, όμως θέλω να πω το εξή ότι οι περισσότερες από τις πρωτοβουλίες αυτές δεν ε, προέρχονται από το ε, γεωργικό τομέα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, όμως σε αυτό το τομέα ήδη ο Επίτροπος ε, είχε προτείνει να διευρύνουμε τις ε, προσπάθειες ε, για τις διεξόδους που έχουν οι γοργοί κυρίως πρέπει να τους χάρη στις τοπικές αγορές μέσω και της οργάνωσης των ε, συνεταιρισμών των αγροτών. Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας βοηθήσει στη μείωση της πετάλης των τροφίμων ε, που πολλές φορές γίνεται στις παραδοσιακές τροφικές αλυσίδες. Επίσης, η αγροτική πολιτική ήδη υποστηρίζει δράσεις, ευαισθητοποίησης στα σχολεία για να προωθηθούν υπεύθυνε και υγιεινές συμπεριφορές κατανάλωση έτσι λοιπόν, ε, ακόμη και αν έχουμε παραμείνει για νομικούς λόγους κυρίως μόνο στο πρόγραμμα της προώθησης βρούτων και λαχανικών στα σχολεία, ε, τώρα αρχίζουμε να θέτουμε, να δίνουμε έμφαση ε, και σε εκπαιδευτικές ενότητες για τα θέματα αυτά. Έχουμε τη σύμπραξη για την καινοτομία στη Γεωργία που προσπαθεί να δημιουργήσει διάφορες μεταξύ της έρευνας ε, και τους πρωταγωνιστές ε, της ε, τροφικής και επιστημιστικής αλυσίδας ε, έτσι λοιπόν ε, ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ε, σε καινοτομίε που θα μειώνουν την σπατάλη των τροφίμων. Αυτά είναι ορισμένα πρωταρχικά στοιχεία σε σχέση με τις δράσεις που είναι ήδη εξελίξει ή που σκοπεύουμε να αναλάβουμε. Φυσικά σημειώσαμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε τις δικές σας ενισφορέ και φυσικά θα ενημερώσουμε και τους συναδέλφους από τις άλλες υπηρεσίες κομισιών σε σχέση με τις προτάσεις που αφορούν ε, τις δικές τους αρμοδιότητες ε, και ήδη ε, θέλουμε εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θεωρούμε ότι η δική σας πρωτοβουλία θα δώσει την απαραίτητη όθηση για να υπάρχει σημαντική πρόοδο σε αυτό το σημαντικό τομέα. Σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη, αλλά η συζήτηση με τον κύριο Σαβίσκη μείωσε το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και έχουμε και τη συνεδρίαση των συντονιστών. Να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Καρόνα για τα καταληκτικά σχόλια και φυσικά θα επανέλθουμε. Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι πετύχαμε τον κύριο στόχο Δηλαδή να στήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό που για πολύ καιρό είχε υποτιμηθεί. Εγώ είμαι πραγματικά ικανοποιημένο από το ότι είχαμε μια τόσο ευρεία συζήτηση και στο εσωτερικό αυτή τη Επιτροπή. Πιστεύω ότι ο κύριος στόχος σε αυτό το πρώτο στάδιο είναι αυτός, δηλαδή να θέσουμε υπό το φως της δημοσιότητας, ε, υπό το φως των προβολέων αυτό το ζήτημα. Ε, όπως ανέφεραν και άλλες συνάδελφοι, γίνεται ένα από τα καθοριστικά στοιχεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία αναπόφευκτα προκαλεί και θα προκαλέσει δυσκολίες διαχείρισης ε, στα επόμενα χρόνια ε, του μεγάλου θέματος των τροφίμων. Έτσι λοιπόν, εγώ περιμένω τις τροπολογίες σας που θα εμπλουτίσουν τη γνωμοδότησή μου και θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε μια πρόταση που θα βρίσκει ω όσο δυνατόν περισσότερους πιο σύμφωνους και που θα μας επιτρέψει να επιβάλλουμε στην Επιτροπή και στα κρατη mail μια συγκεκριμένη στρατηγική για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για να καταστήσουμε την Ευρώπη όπου μαζί με τη ΣΥΠΑ υπάρχουν μεγαλύτερες πατάρες αυτή τη στιγμή για να καταστήσουμε λοιπόν την Ευρώπη μια περιοχή όπου θα, η οποία θα παρεμβαίνει όσο δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη επιστημιστική ασφάλεια. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα τη συζήτηση και θα περάσουμε ε, τώρα στο σημείο 13 σε ό,τι αφορά τον τριμερή διάλογο. Η Μπρίτα. Ε, Σύντομα, να σας φέρω ευχάριστα νέα. 27 Ιουνίου συμφωνήσαμε στην πρώτη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου για την προαιρετική διαφοροποίηση άμεσων πληρωμών. Υπήρχε μία μικρή αλλαγή στο άρθρο 6 παράγραφος 2 για συμβουλευτική διαδικασία. Έγινε διαδικασία εξέτασης και εάν μπορέσουμε να το στηρίξουμε νομίζω στην Ολομέλεια θα έχουμε μία από τις πρώτες συμφωνίας τριμερούς διαλόγου που θα, πάει, θα ολοκληρωθεί στην πρώτη ανάγνωση. Αυτά και ευχαριστώ. Πολύ ωραία, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα ακολουθήσουμε τι ενδείξει τη ΠΛΙΤΑ. Σα ενημερώνω ότι η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα θα είναι στι 30 Αυγούστου. Καλέ διακοπέ λοιπόν σε όλου. Παρακαλώ συντονιστέ να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί θα ακολουθήσει συνεδρίαση των συντονιστών. Και φυσικά να ευχηθώ καλές διακοπές στους υπόλοιπους, θα τα πούμε σύντομα. Και σας παρακαλώ κατευθύντε προς την έξοδο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, 12 και μισή πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ε, ε, ε.